Υπότιτλοι Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer notre euh, réunion en adaptant notre... Θα ήθελα να ξεκινήσω τροποποιώντας ε, την ημερήσια διάταξή μας ε, για την αυριανή μα συνεδρίαση τη 17 η Μαρτίου. Θα αρχίσουμε στις 3.30 το απόγευμα και όχι στις 3 όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη το για να ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα του Επιτρόπου Πίμπαλξ, ο οποίος θα μπορέσει να έρθει στις 5 το απόγευμα αύριο και θα σας το ξαναπώ αύριο το απόγευμα. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και την ελαφρά τροποποίηση. Αν δεν υπάρχουν, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Θα ήθελα επίση να σας ενημερώσω ότι η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οργανώνει μία ακρόαση με τίτλο από την διπλωματία της αντίδρασης στην, διπλωματία της πρόληψης. Ο κύριος Ντόμσκης ε, θα εκπροσωπήσει την ε, δική μας επιτροπή. Όλοι οι ευρωβουλευτές είναι ευπρόσδεκτοι. 9 με 11.30 στην αίθουσα ε, 3ε2 στην Πέμπτη. Ναι, θα ήθελα να πω ότι αύριο είναι St. Patrick's Day για μας. Και θα μας καλέσετε για whisky, ελπίζω. Δεν έχουμε ερωτήσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα περάσουμε στην ψηφοφορία για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Περάσουμε στην ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση της Κατρίν Γκρέζ το πλαίσιο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Πρέπει να το να ξανακάνουμε τη ψηφορία γιατί δεν είναι πολύ σαφές το αποτέλεσμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Καταπίπτει και αυτή. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία από τον κύριο Φίσας. Υπέρ. Κατά. Κίσε. Αποχές. Εγκρίνεται. Σε κομπρομί 2. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αμάντμα 14. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Υπάρχει μια αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Οπότε δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Oui, 18. Donc, euh, c'est ça, c'est 18 en vote. Ouais. Donc, amendement 10. Τροπολογία 18. Υπέρ. Non, non, la 18 tombe aussi, hein. Pardon. Oui. False, if 17 is adopted. It's 16, which is adopted. This one was adopted. 17? No. Ah, sorry. Shall we? I'm sorry. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, από την αρχή. Τροπολογία 18, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 5. Υπέρ. Υπάρχει αντίρρηση. Οπότε δεν την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. On peut compter. Mais vous n'avez pas compté. Bon, alors on recommence. Άλλη μια φορά. Υπέρ. Για την τροπολογία 21 πάντα. Υπέρ. Qui sont contre Κατά. αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Καταπίπτει. Τροπολογία 26. Υπέρ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Λέει ότι καταπίπτει αν η τροπολογία 21 εγκρίνεται. L'amendement Εγκρίθηκε η τροπολογία 21. 12 προς 11. Αυτό σημαίνει ότι η συμβιβαστική 4 καταπίπτει. Συγγνώμη να κάνω. Θέλω ένα διαδικαστικό να θέσω. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τη διαδικασία. Για την πρώτη παράγραφο ψηφίσαμε πρώτο το συμβιβασμό. Ψηφίσαμε πρώτα τη συμβιβαστική 1 και μετά την τροπολογία 1. Γιατί δεν κάνουμε και το ίδιο και στην παράγραφο αυτή που ψηφίζουμε τώρα. Ναι. Alors, <clears throat> cela fait l'objet d'une étude de la part du secrétariat. Κοιτάξτε, το μελέτησε αυτό η γραμματεία. Έχω εδώ τον κανόνα 160 που λέει Διακόπτη η πρόεδρος. Όταν προτείνεται μια συμβιβαστική τροπολογία στην Επιτροπή, η συμβιβαστική τροπολογία έχει προτεραιότητα στην ψηφοφορία. Αλλά ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τις ψηφοφορίες ε, στις επιτροπές ε, βάσει του κανόνα 196 που αναφέρει ότι οι τροπολογίες ε, ότι οι κανόνες που ισχύουν για την Ολομέλεια δεν ισχύουν υποχρεωτικά για την ε, ψηφοφορία στις επιτροπές. Έχουμε λοιπόν και τον κανόνα 160 και τον 161, αλλά δεν αναφέρεται στον κατάλογο ε, των κανόνων που ισχύουν και για τις δύο περιπτώσεις. Οπότε αυτός είναι ο κανονισμός ε, που ισχύει. Μάλιστα, τότε μήπως μπορούμε να επαληθεύσουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 21. Ναι, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, για την τροπολογία 21 ψηφίσαμε δύο φορές. Ε, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Επειδή ήταν ε, πολύ τσιματσίμα η ψηφοφορία, μήπως δεν είναι πολύ καλή ιδέα να επαληθεύσουμε πάλι μια ψηφοφορία που με τόσο τσίμα τσίμα τρόπο πέρασε. Ναι, το ξανακάναμε, δύο φορές το ψηφίσαμε λέει η Πρόεδρος, 12 υπέρ 11 κατά. Οπότε έχει εγκριθεί η τροπολογία 21 και τέλος. Ωραία. Συνεχίζουμε με την 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Δώδεκα. Κατά. Αποχές.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 Nous maintenant le plaisir d'accueillir. Έχουμε τώρα την ε, ικανοποίηση να καλωσορίσουμε την κυρία Κριστέλινα Γεωργίευα, Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων. Ε, πρώτη φορά η κυρία Γεωργίευα παρουσιάζεται εδώ στην Επιτροπή μας ε, από την κρασί τη, από όταν έλαβε τα καθήκοντά τη το Φεβρουάριο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάληψη των καθηκόντων της και την ευχαριστούμε για την παρουσία της. Η κυρία Γεωργίευα θα μας ε, ε, γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της πρόσφατης αποστολής της στην ΑΕΤ και θα μας μιλήσει για τις μεγάλες προτεραιότητες των επόμενων μηνών. Έχετε το λόγο κύριε Γεωργίευα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έψαχνα την καλλική λέξη. Η συγκητή συγχύτρια λέει κυρία Γεωργίευα. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία να επανέρχομαι εδώ ως ε, Επίτροπος που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της και σας, ευχαριστούμε, και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια της ακρόσης και τη διαδικασία του διορισμού μου. Όπως είπα, όταν ε, πρωτοσυναντηθήκαμε είναι τιμή αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη να είμαι Επίτροπος για τον χαρτοφυλάκιο Διεθνής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοηθείας και Αντιμετώπιση των Κρίσεων ο πρώτος ε, μήνας ε, ε, της θητείας μου, τη και των καθηκόντων μου, το έδειξαν αυτό, καθώς είχαμε μία σειρά φυσικών καταστροφών μετά την ΑΕΤ, το σεισμό της ΑΕΤ τον Ιανουάριο, είχαμε και καταστροφές σεισμού στην Τουρκία και στη Χιλή και καταιγίδε και φυσικά έχουμε και τις κρίσεις στο Σουδάν, στη Σομαλία, στο Αφγανιστάν, στη Μέση Ανατολή, για να αναφέρω μερικές. Σήμερα θα ήθελα να σας αναφέρω ποια είναι η εμπειρία που αποκόμισα από την Αϊτή και τη Χιλή. Να σας παρουσιάσω λεπτομερέστερα τις προτεραιότητές μου και κατόπιν να ακούσω τις δικές σας συμβουλές και σκέψεις. Και ε, ε, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να καθορίσουμε τους ευρύς προσανατολισμούς και να έχω το δικό σας feedback, τη δική σας ανάδραση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τι εργασίε μα στον ορθόδρομο, γιατί ήταν και είναι στην κορφή τη ατζέντα μου, όπω αναφέρει η κυρία Ζολή, πριν δύο εβδομάδε ε, μετέβη στην ΑΕΤ και είδα τις καταστροφές και το πόσο τα δεινά των ανθρώπων, είδα όμως και την αξιοπρέπεια του λαού της Αιτής ε, και τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει η διεθνή κοινότητα για να προσφέρει βοήθεια. Επίσης ε, είδα ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ εδώ με υπευθυνότητα να πω ότι δράσαμε αποτελεσματικά και ταχύτατα από την πλευρά της Κομισιόν. Εμείς ε, ε χάρη και στο Κοινοβούλιο ως Δημοσιονομική Αρχή ενεργοποίησαμε περίπου 100, 120 εκατομμύρια ευρώ τέσσερις φορές το ποσό που κατανέμηθηκε, που εκπονήθηκε συγγνώμη για την ε, έναρξη της καταστροφής. Επίσης, συντονίσαμε τη βοήθεια από 25 κράτη-μέλη και είναι δίκαιο να πούμε ότι συνολικά ε, ε, δώσαμε τη σωστή βοήθεια, τη σωστή χρονική στιγμή και ε, έτσι ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Είδα την κατάσταση των νοσοκομείων, είδα την παροχή τροφίμων και πραγματικά με συγκίνησε μια εικόνα που είδα ενός μικρού παιδιού το οποίο σώθηκε γιατί πραγματικά αποφασίστηκε ε, η ομάδα που αρρωγής που είχε σταλεί να μείνει μία μέρα παραπάνω για να με υποδεχτούν εμένα και αφού ε, επισκέφθηκα τις περιοχές που πλήγησαν περισσότερο, θα ήθελα να σας αναφέρω πέντε κυρίες παρατηρήσεις ή διδάγματα από το ταξίδι. Καταρχήν, Σήμερα οι βασικές ανθρωπιστικές ε, ανάγκες ε, είναι ε, τα τρόφιμα, το νερό και κάποια μορφή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φυσικά στέγαση. Κάποιες από αυτές καλύπτονται, κάποιες από αυτές τις ανάγκες, όμως εξακολουθούμε να είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί θα έρθουν και και υπάρχουν κάποιες ε, πραγματικές ανθρωπιστικές ανάγκες που πρέπει να επιληθούν κυρίως ότι φορά τη στέγαση, ε, το είναι διατροφή, την υγιεινή ε, και διατροφή κυρίως για τις πιο ευπαθείς ομάδες και η βοήθειά μας των Ελλήνων και Ευρώ θα επικεντρωθεί σε αυτό. Επίσης, πρέπει ε, να λάβουμε μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ε, όπως ε, να έχουμε αποθήκευση σε θέματα σε τρόφιμα και πρέπει να σκεφτούμε και τη Δομικανή Δημοκρατία, πρέπει να σκεφτούμε την ίσω το σύνολό τη. Ε, και ε, επίση ε, πρέπει και εκεί να φροντίσουμε να υπάρχουν προμήθεια σε τρόφιμα γιατί ξέρετε πολλές φορές ότι υπάρχουν φυσικές καταστροφές και υπάρχει πρόβλεψη ότι μπορεί να χτυπηθούν από φυσικές, μπορεί να χτυπηθεί από φυσικέ καταστροφέ στην Τρίτον, η ανθρωπιστική βοήθεια εξαρτάται από το να διατηρούμε βασική επιμελητία ε, και τι υποδομέ σε κατάσταση λειτουργία. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να χρειάζονται ε, στρατιωτικέ δυνάμει ε, και ξέρουμε ότι υπάρχει κινητοποίηση των Καναδών. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μειώνουν την στρατιωτική του υποστήριξη. σω πρέπει να σκεφτούμε εμεί λοιπόν από την πλευρά των κρατών μελών λοιπόν ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για θέματα βασικών υποδομών. Τέταρτο, και θέλω να το τονίσω αυτό ολόψυχα, θεωρώ ότι αυτό είναι μέγιστη προτεραιότητα για μας. Ε, εμείς ε, τα πήγαμε καλά στην παράδοση, αλλά δεν τα πήγαμε καλά σε ό,τι αφορά την προβολή και υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα κράτη-μέλη και τα μέσα μαζική ενημέρωση να εργαστούν για να ε, ενημερώνουν καλύτερα για τη συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είχα μαζί μου ένα σημειωματάριο, γιατί ήθελα να σημειώνω πόσε φορέ και πού ε, βλέπα την Ευρωπαϊκή Συμβολή και τελικά τέσσερι φορέ το είδα. Δεν χρειαζόμουν να κάνω σημειωματάριο. και είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ε, είναι εδώ μια ένα πρόβλημα όταν θέλουμε οι φορολογούμενοι μας να γνωρίζουν ότι εμείς συνεισφέρουμε ε, για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και πέμπτον, πρέπει να διασφαλίσουμε σύνδεσμο μεταξύ της ε, ανακούφισης, της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Και τι κάνουμε από την ανθρωπιστική προσκοπία, να προωθήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, όχι στο ε, Πόρτο πράγμα, να μην τη συγκεντρώσουμε εκεί, αλλά να την ε, διανύμουμε σε όλοι. Ε, τη χώρα, στο Λόγκαν και σε άλλες ε, περιοχές, ε, εκεί όπου οι άνθρωποι μετακινούνται για να ζήσουν με τους συγγενείς τους αλλά οι συνθήκε είναι πάρα πολύ ε, άσχημε, Υπάρχει πολύ φτώχεια και μιλάμε για 500-600 χιλιάδες άτομα ε, μπορεί να επιστρέψουν στο Πορτοπράνς και ήδη η δύσκολη κατάσταση να γίνει πελητριστική. Και μέχρι τον Ιούνιο θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις εργασία και να ε, δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια, όχι αποκλειστικά στο, αλλά εκεί όπου μετακινούνται οι άνθρωποι. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία σημαντικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη της χώρας. Μία ακόμη πτυχή. Μπορούμε να συνδέσουμε την βοήθεια με την ανάπτυξη και αν συμπεριλάβουμε στις ανθρωπιστικές ε, πρωτοβουλίες κάποια προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, και Επίσης, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και ακολουθεί τα βήματα των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολύ συνεργασία, καλή συνεργασία με τον Επίτροπο Πίμπαλξ μαζί υπό την ηγεσία της κυρίας Άστον θα μεταβούμε σε μια συνδιάσκεψη στις 31 Μαρτίου για την ανοικοδόμηση της Αιτή και νομίζω ότι αυτή η συνδιάσκεψη θα μας βοηθήσει στο να σκεφτούμε πώς θα οικοδομήσουμε την ΑΕΤ, όχι μόνο όμως από τη σκοπιά της ανοικοδόμησης μετά το σεισμό, αλλά και πώς θα ε, διορθώσουμε όλες αυτές τις δεκαετίες της κακής διακυβέρνησης. Ο σεισμός είναι κάτι τρομερό, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της IT. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της IT είναι αυτή η κληρονομιά της υποανάπτυξης που υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Και αυτό το θέμα του να συνδέσουμε την ανακούφιση, την ανθρωπιστική βοήθεια με την ανάπτυξη ε, θα το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά και εγώ και ο Επίτροπος Πίλβαξ και ως θέμα χάραξης πολιτικής αλλά και ως επιχειρησιακό ζήτημα σε επίπεδο χώρες. Να πω τώρα δυο για τη Χιλή. μας ε, σε αυτή την αίθουσα βίωσαν ε, τον σεισμό του 7,2 Ρίχτερ. Ο αντίκτυπος ε, στις, στις περιοχές που πλήγησαν περισσότερο είναι πραγματικά τεράστιος. Υπάρχουν χωριά που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά από το τσουνάμι, όμως η χιλίδες στο σεισμό 8,8 ε, βαθμό της κλίμακας Ρίκτερ ε, και περίπου 500 άτομα πέθαναν στη Χιλή και οι περισσότεροι από το τσουνάμι, όχι από το σεισμό, ενώ είχαμε 220.000 άτομα που σκοτώθηκαν στην Αϊτή ε, λόγω του σεισμού. Γιατί η Χιλή έχει επενδύσει δεόντως στα ορθά πρόκτυπα των κτηρίων, τα οποία σώζουν ζωές και έχει επενδύσει στην προστασία από τους σεισμού και η ταχεία μα ε, ανταπόκριση στη Χιλή πραγματικά εκτιμήθηκε από το λαό τη Χιλής ο ε, οποίος ε, πραγματικά γνώρισε εκεί νοσοκομιακή περίθαλψη, προσωρινή στέγαση, μηχανικές γέφυρες και επίσης ε, εκτίμησαν και οι πρεσβευτές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χιλή που είπαν ότι όταν η Κομισιόν μπορεί να δράσει άμεσα τότε αυτό βελτιώνει σημαντικά την φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμω στη Χιλή ήταν σαφές το τι έπρεπε να γίνει. Κυρίω σε ό,τι αφορά τα συστήματα επιφυλακής. Ε, τα το σύστημα επιφυλακή για το τσουνάμι σε εθνικό επίπεδο ε, μπορεί να είναι αντικείμενο διαχείρισης και σε τοπικό επίπεδο. αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν χωριά όπου πέθαναν άνθρωποι από το τσουνάμι και άλλα χωριά τα οποία χτυπήθηκαν λιγότερο. Έτσι λοιπόν, εκεί όπου λειτουργήσαν τα συστήματα επιφυλακής, έσωσαν ανθρώπινες ζωές. Αυτέ οι δύο τραγωδίες με οδηγούν στο κύριο θέμα που θέλω να αναφέρω σήμερα ότι ε, ε, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εντολή για αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο είναι να προετοιμάσουμε τις ικανότητες ε, ετοιμότητας και να μπορούμε ταχύτατα να ανταποκριθούμε στις καταστροφές ανεξάρτητα από τις ε, τοπικές συνθήκες να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ε, υφιστάμενη ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έτσι ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ταχύτερα όταν χτυπήσει η επόμενη καταστροφή στο ψήφισμα που πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υιοθετήθηκε γέρο και εμείς φυσικά θα σκεφτούμε δεόντως επί των θεμάτων αυτών. Έχω υψηλές φιλοδοξίες ε, για το θέμα αυτό και θα εργαστώ πάρα πολύ εντατικά για να ενισχύσω τους ε, φορείς ε, ετοιμότητας και ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συναδέλφου Σεσίλια Μάλστρομ και Κάθι Άστον και επίσης θα συνεργαστούμε στενά και με τον Επίτροπο Πίμπερξ για να ε, έχουμε μία διάσταση πρόληψης των κινδύνων η οποία θα συνάδει και με την κλιματική αλλαγή. Ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή βάση για να πετύχουμε το στόχο αυτό αν λάβουμε υπόψη και τις αλλαγές, συγγνώμη, και τις πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές. Τώρα να σας πω ποια είναι η ατζέντα μου για τις υπόλοιπους επόμενους μήνες. Έχουμε την ενδιάμεση επισκόπηση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό θα γίνει σε διάλογο μαζί σας, αλλά και με άλλους εταίρους. Μέχρι είναι μια ευκαιρία κατά τη διάρκεια της αναθεώρηση να συνεισφέρουμε για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και το συντονισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση αυτό αποτελεί ευκαιρία να αυξήσουμε και να ενδυναμώσουμε το ρόλο μας στο να βελτιώσουμε την παγκόσμια ανθρωπιστική διακυβέρνηση. Θα πρέπει ε, το οικονομικό μας βάρος να συνάδει με το πολιτικό μας βάρος στα θέματα αυτά. Η δική σας έκθεση θα συνεισφέρει τα μάλα στην εργασία αυτή, όπως ε, και οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα αύριο μετέρους εδώ στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Σκοπεύω να υιοθετήσω μια πολιτική δήλωση το φθινόπωρο και ε, να ε, παρουσιάσω και το πρόγραμμά μας μέχρι το 2013. Δεύτερον, θα εφαρμόσω την εντολή ε, για να έχουμε το 2011 το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα ε, μέχρι το τέλη του 2010 θα αναπτύξουμε μια σχετική πρόταση. Θα σκεφτούμε τα διδάγματα που έχουν αποκομιστεί από τις υφιστάμενες προκλήσεις ε, και τα προβλήματα για την χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα λάβουμε όψη το κόστος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα ήδη. Ε, ε θεωρούμε, οργανώνουμε μάλλον μία διαβούλευση όπου θα συμμετέχουν όλοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να έχουμε μία ισχυρή πλατφόρμα προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή ευρωπαϊκές αξίες που θα σέβεται τα ε, επαγγελματικά πρότυπα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ε, θα σέβεται και τους νέους ανθρώπους. Ε, σε σχέση με τη συνεργασία μου με την Κάθριαν Άστον, θα έχουμε μια διευρυμένη συζήτηση για τη ταχεία στρατιωτική δράση. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς σε μια περίπτωση καταστροφής αντιδρούμε ε, και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε όσο δυνατόν καλύτερα όλα τα μέσα και τα στρατιωτικά μέσα και να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα σε όλο τον κόσμο. Υπήρχε θετική πρόοδος ε, τα τελευταία χρόνια και έχουμε και διδάγματα από την επιχείρηση U4 στο Τσάντ θα οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό δόγμα και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους ε, Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας. Επίσης, θα προωθήσουμε το σεβασμό του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Ευρωπιστικού Δικαίου. Εμείς ε, θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, θέλω να δεσμευτώ στις δύο αρχές. συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη ε, και με τους ε, υπόλοιπους εταίρους μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Έχετε το λόγο ο κύριος Μαρτίνες, πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να καταστώ μάρτυρας για τη δράση της Επιτρόπου στην πρόσφατη επίσκεψή της στη Χιλή. Όπως είπε και η κυρία Γεωργίευα, συμπέσαμε εκεί, εγώ εκπροσωπώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Γεωργίευα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να πω στους συναδέλφους το εξή. Το να κάνουμε μια θετική κριτική οποιασδήποτε δράση ε, της Κομισιόν ε, μας ε, δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε και κριτική. Όμως η δράση της κυρίας Γεωργίευα ήταν εξαιρετική κατά την άποψή μου και ακολούθησε τις ε, εξαιρετικές εντυπώσεις ε, που αποκομίσαμε οι περισσότεροι από εμά τη στιγμή της ακρόασης της ενώπιον ε, στην Επιτροπή, της Επιτροπής μας. Όταν παρουσίασε την υποψηφιότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επίτροπος. Βέβαια, θα ήθελα να φερθώ και στι θετικέ εντυπώσει που αποκομίσαμε από τι συνεδριάσεις που είχε και η κυρία Γεωργίευα με του πρεσβευτέ όλων των κρατών μελών. Και σήμερα και με τη συνάντηση που είχε με το σημερινό πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χιλή. Η κυρία Γεωργίβα μας εξήγησε με πολλές λεπτομέρειες και μάλιστα με περισσότερες λεπτομέρειες από τη σήμερα γιατί τότε υπήρχε πολλής χρόνος ε, και ήταν και μικρότερη σύνθεση της ομάδας. Μας εξήγησε ποια είναι την αποστολή της λοιπόν αλλά εμείς την προηγούμενη μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, μπορέσαμε να διαβάσουμε διάφορες ε, πληροφορίες και είδαμε και στην τηλεόραση ποιος ήταν ο αντίκτυπος της δράσης της στην ε, δημόσια στην κοινή γνώμη της Χιλής και μάλιστα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο λαός στη Χιλή αυτή τη στιγμή έχει πληγεί ιδιαίτερα από το σεισμό. Έτσι λοιπόν ε, όταν ε, κάποιος ε, εκπροσωπεί και μιλάει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο σε τέτοιες καταστάσεις η κυρία Γεωργίευα μας ε, εξέθεσε σήμερα το ρόλο που διαδραμάτισε εκεί. Εγώ όμως θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι συνάντησε και τους πρεσβευτές και τους ε, παρότρινε να συντονιστούν στη δράση τους, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της ε, Επιτροπής. Και ουσιαστικά τους παρότρινε έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή στη δράση όλων ε, των πρεσβευτών των κρατών μελών. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι με κάποια έκπληξη εγώ άκουσα την ανησυχία κάποιων ε, πρεσβευτών οι οποίοι ε, είπαν ότι ποτέ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια μάλλον, ε, κάποιος Ευρωπαϊκός Επίτροπος δεν έχει επισκεφτεί τη Χιλή, όπως και τη Βενεζουέλα άλλωστε. Και έλαβα τέτοιε πληροφορίες πριν κάποιες εβδομάδες όταν εγώ επισκέφτηκα εκείνη τη χώρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό συμπέρασμα που εξάγεται από την αποστολή της κυρίας Γεωργίευα ότι η Επιτροπή μας πρέπει να επισκέπτονται τις χώρες που είναι εταίροι μας και να μην το πράττουμε αυτό μόνο όταν λαμβάνει η χώρα κάποια καταστροφή αλλά και υπό κανονικές συνθήκες προκειμένου να εξηφαίνουμε πιο στενές σχέσεις. Λεχθέντων αυτό να κάνω και κάποια σχόλια για τις εντυπώσεις που αποκομίσα και εγώ από τη Χιλή ως αντιπρόεδρος και ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, η εντύπωση μου ήταν ότι στην περίπτωση, η περίπτωση της Χιλής και η περίπτωση της ΑΙΤΙΣ ε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια χώρα όπως η Χιλή όπου λειτουργεί το κράτος δικαίου και υπάρχει ουσιαστικός ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ε, εμπειρία και υπάρχουν και ε, Παρκή ανθρώπινη και οικονομική πόρη προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει από μόνη της τέτοιες καταστροφές όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση, στην κατάσταση λοιπόν της Χιλής πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ε, μιλάμε για μια χώρα στην οποία το βιωτικό επίπεδο είναι πιο υψηλό από κάποια 8-9 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να αποφύγουμε τη σύγχυση, να ε, θεωρούμε ότι η ΑΕΤ και η Χιλή είναι στην ίδια κατάσταση. Σε συζητήσεις ε, που είχα εγώ με άλλους χιλιανούς, ε, Πριτάνη στο Πνευστημίο κτλ, μου είπαν ότι ε, πραγματικά ε, αισθάνονται άσχημα να λένε σε κάποιους από τους δωρητές «Κοιτάξτε, εμείς στην πραγματικότητα δεν το χρειαζόμαστε αυτό». Όταν ε, γίνεται μια τέτοια καταστροφή, ε, λόγου χάρη μπορεί μια χώρα να προτείνει να στείλει πυροσβέστες όμως ε, στην ε, Χιλή υπάρχουν 2.000 πυροσβέστες γιατί έχουν πάρα πολλούς σεισμούς το χρόνο και έτσι λοιπόν είχαν ε, σταλεί λόγου χάρη όταν ε, έγινε η καταστροφή στην Ιταλία, είχαν σταλεί πυροσβέστες γιατί στην Ιταλία δεν υπάρχουν ε, τέτοιοι πόροι, όμως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν γίνεται από φέτος, πρόκειται για μια αναπτυγμένη χώρα, για μια χώρα η οποία διαθέτει ανθρώπους με υψηλά προσόντα και ο ίδιο συνεργασία είναι αυτό που παρουσίασε η κυρία Γεωργίευα, δηλαδή να μπορούμε εμεί να παρεμβαίνουμε όπω όταν παρεμβαίνουμε αν υπάρχει παρόμοια καταστροφή στην Ισπανία, στην Ιταλία ή στη Γερμανία. Δεν είναι η καταστροφή ίδια όπω στην ΑΕΤ, όπου ε, η ανοικοδόμηση τη χώρα και η ανθρωπιστική βοήθεια ε, καταστούν απαραίτητη την παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Εγώ νομίζω ότι η ελεγγύη που εκφράστηκε ουσιαστικά παγιώνει και κάποιες αδερφικές ε, σχέσεις που ήδη Και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά εμένα μου δόθηκε εκεί μία αίσθηση ασφάλειας γιατί ε, εμείς ε, ήμασταν πάρα πολύ ήσυχοι εκεί όταν έγινε ο σεισμός απλώς καθίσαμε ήρεμοι ήρεμοι στην καρέκλα μας ε, και περιμέναμε <laughs> και είναι 20, 20 δευτερόλεπτα κράτησε η κυρία Επίτροπος πραγματικά ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μοιάζαμε σαν αυτά τα μηχανήματα που τους ρίχνει σε ένα ευρώ και τρέμουν κάπως. Ε, Πάντω ε, ήθελα να αναφέρω αυτή την εμπειρία μου. Πάντω ευχαριστώ Πρόεδρε και συγχαρητήρια κυρία Επίτροπε για τη δράση σα στη συγκεκριμένη περίπτωση και ελπίζω να επαναληφθεί σε όλε τι περιπτώσει. Ο κύριο Μπέρμαν παρακαλώ. Oui. Mevrouw de commissaris, dank u Κύριε Επίτροπε, ε, σας ε, ευχαριστώ θερμά για αυτή την ε, τόσο σύντομη και ξεκάθαρη παρέμβασή σας και με πολύ δυναμισμό μάλιστα. Θα ήθελα όμως να σας ερωτήσω κάτι. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα περιουσιακά θέματα. Δηλαδή υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι και απολύτως απαραίτητο. Ε, θα πρέπει αυτό το στοιχείο να ενισχυθεί περισσότερο από την επικοινωνία. Ε, όμως η επικοινωνία μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω μόνο εφόσον υπάρχει γνώση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μία συζήτηση ε, σχετικά με την πρόληψη της κρίσης, την ομάδα κρούσης. Ε, πώς θα διαρθρωθεί αυτή. Υπάρχουν κάποιες ε, αμφιβολίες ε, στο Συμβούλιο για το ότι αυτή η ομάδα κρούσης δεν θα είναι τόσο σαφής και αυτό το επικρίνουν πολλοί. Μπορεί κανείς να πει ότι θα μπορούσε να είναι μια οργάνωση στην οποία διαθέτουν όλα τα κρατη ομάδες ε, επιμελητίας, γιατρών ε, και πολλών άλλων επαγγελματιών, έτσι ώστε η ομάδα αυτή να είναι διαθέσιμη για την περίπτωση που είναι χρήσιμη. Ε, η ομάδα αυτή θα μπορούσε να είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών και αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ε, χαλαρή και πολύ πιο ευέλικτη. Ε, Παραδείγματο χάρη μπορεί κανείς ε, να σκεφτεί και να αποφασίζει κάθε φορά κατά περίπτωση ποια χώρα θα έχει την, την εξουσία, ποια θα έχει το συντονισμό μιας τέτοιας ομάδας. Αυτό θα κρίνεται από τον χώρο όπου προκύπτει η καταστροφή Μπορούν να παίξουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα ρόλο για να κρίνετε καλύτερα ή κάθε φορά να κρίνετε οι ανάγκες που υπάρχουν. Σας, ήθελα να σας ρωτήσω όμως, αυτές οι κρίσεις και αυτή την ομάδα κρούσης, ε, πώς ακριβώς κρίνετε τις ε, σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ο κύριος παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε αν ήταν όλα τόσο σαφή όσο ο λόγος της κυρίας Γεωργίευα θα είχαμε πολύ λιγότερα ερωτήματα να θέτουμε σε επίπεδο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σε σχέση με την κατανομή εργαζιών μεταξύ της ε, κυρίας Άστον και της Επιτροπής. Ελπίζω ότι η σαφήνεια την οποία επιδείξατε να γίνει ιός που θα προσβάλλει όλα τα ε, όργανα της ε, διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω αφορά την ΑΕΤ. Πήγατε εκεί και είχατε τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με τις πολιτικές αρχές ε, της χώρας. Κρίνετε την ικανότητα των πολιτικών αρχών της ΑΕΤ ως επαρκή, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για συνεργασία. Υπάρχει η απαραίτητη δυνατότητα ώστε η ΑΙΤΗ από τώρα να συμμετέχει στην ανοικοδόμηση, στην ανάπτυξη και στην πλήρη αποκατάσταση της χώρας. Γιατί είναι γεγονός ότι την ε, ε, επόμενη μέρα των, ε, του σεισμού ε, είναι γεγονός ότι και σε πολιτική κατάσταση επλήγει ιδιαίτερο η χώρα και υπήρξε ιδιαίτερη αναστάτωση, εν μέρει έχει αποκατασταθεί αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, και είναι κάτι το οποίο μεταγενέστερα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα, Πρόκειται για την ύπαρξη ενός συστήματος αμοιβαιότητας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των χωρών στις οποίες υπάρχει άμεση ανθρωπιστική παρέμβαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει σημασία ε, σε ποια μορφή γίνεται αυτό. Απλώς θα ήθελα να ρωτήσω ποιος, πώς πηγαίνουν τα πράγματα σε σχέση με το θέμα αυτό. Κυρία Γεωργίευα, έχετε το λόγο για να απαντήσετε τις πρώτες αυτές τις ερωτήσεις. Uh, thank you very... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που προσφέρετε σε μένα και στους ε, συνεργάτες μου που ε, συνεργάζονται μαζί μου στις διάφορες χώρες που παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ε, υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει μεγάλη απήχηση στις χώρες στις οποίες ε, δραστηριοποιείται. Να τοποθετηθώ σε τρία θέματα επιθυμώ. Πρώτον, όσον αφορά στο ότι σε αυτά που είπε ο κύριος Μαρτίνες για τον σεισμό για την εμπειρία που διαθέτουμε στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσσουμε ε, τις σωστές δυνάμεις ε, στο σωστό χρόνο και στο σωστό χώρο και να μην ε, ισχυριζόμαστε βέβαια ότι η Ευρώπη είναι καλύτερη από άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί στον σεισμό ειδικά η Χιλή διαθέτει ένα εντυπωσιακό δυναμικό και μάλιστα ένας από τους ε, συνεργάτες μου είπε Κάποιος με ρώτησε αν έχω ε, blog ή Twitter. Κάποιος λοιπόν από τους ε, συνεργάτες μου είπε ότι αν πρόκειται να βρεθεί σε ένα σεισμό, καλύτερα βρεθεί στη Χιλή, όχι στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει το ίδιο δυναμικό. Ίσως στην Τουρκία τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα, να είναι καλύτερα προετοιμασμένη χώρα. Όμως εδώ αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι χωρίς ε, συντονισμό δεν θα μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που προσφέρουμε την ώρα της ανάγκης πράγματι είναι και το απολύτως απαραίτητο. Φτάνω λοιπόν ε, σε αυτά που είπαν ο κύριος Μπέρμαν και ο κύριος Γκιόνης, δηλαδή τι ακριβώς προγραμματίζουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το επίπεδο του συντονισμού και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Σήμερα βρισκόμαστε στο εξής ε, σημείο. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, διαφορετικές απόψεις και θα έλεγα μάλιστα ορισμένα κράτη-μέλη διαφοροποιούνται σημαντικά στο πώς ακριβώς προβλέπουν τη βελτίωση του συντονισμού. Ε, έτσι λοιπόν, για να είναι η συζήτηση λίγο πιο απλή, θα έλεγα ότι υπάρχουν για μας τρεις δυνατότητες για να προχωρήσουμε. Η μία είναι να μην κάνουμε τίποτα, δηλαδή να έχουμε αυτό που έχουμε, ε, να παραμένουμε στην καλή συνεργασία και τον καλό συντονισμό, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον συντονισμό και παραμένουμε όμως εκεί. Ε, δεύτερον, να είμαστε καλύτερη στο συντονισμό, πιο αποτελεσματική, αλλά μέχρι εκεί. Το δεύτερο, να μπορέσουμε να συστήσουμε ένα κεφάλαιο κοινό για όλους μας, ε, αποτελεσματικό από σε κόστος ωφέλους, έτσι ώστε αυτό είτε να υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος, είτε ε, σε μια κοινή δεξαμενή υπό τον έλεγχο της Κομισιόν, υπό την κυδαιμονία της Κομισιόν, για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει σε περίπτωση ε, καταστροφής. Το άλλο είναι ότι μπορούμε ε, να προχωρήσουμε ένα βήμα περαιτέρω προς αυτό που προτείνει η έκθεση Μπαρνιέ, δηλαδή μια γνήσια υπηρεσία πολιτικής προστασίας η οποία να χρηματοδοτείται από όλα τα κράτη-μέλη και να είναι στην υπηρεσία όλων για το κοινό καλό. Το έχω αυτό ε, συζητήσει με πολλά κρατημέλη και δεν έχω αυταπάτες, ε, δεν θα είναι εύκολο να συμφωνήσει κανείς πάνω σε όλα αυτά. Όμως ε, είμαι απόλυτα αποφασισμένη να πίσω τα κρατημέλη, να εξετάσουν αυτές τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν και έτσι τα κράτη-μέλη να καταλήξουν ε, σε ένα καλύτερο επίπεδο από αυτήν την επιλογή που είναι του ε, δύο και τίποτα παραπάνω. Αυτή δεν είναι και η καλύτερη. Ένα παράδειγμα να σας αναφέρω. Στη Χιλή είδα ένα από τα ε, πιλωτικά προγράμματα επιτόπου, ένα πρόγραμμα που να μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε 24 ώρες ανεξάρτητα από τη χώρα που επικρατεί στη χώρα, από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Με άλλα λόγια δηλαδή, ε, δεν ε, περιορίζει τις δυνατότητες της χώρας τη στιγμή της ε, κρίσης. Αυτό ζυγίζει 560 κιλά και με τον τρόπο αυτό τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να στείλουν μεμονωμένες αποστολές γιατί βεβαίως ε, προσφέρουν ένα κοινό καλό για όλους μας. Νομίζω λοιπόν ότι το να το να σε μια καλύτερη, ε, έναν καλύτερο συντονισμό και να βελτιώσουμε την συνεργασία των κρατών μελών, αυτό είναι απολύτω απαραίτητο. Γιατί η τάση είναι σαφή. Οι καταστροφέ είναι πολύ πιο συχνέ, ε, πολύ πιο οξύε ανά τον κόσμο. Ε, έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα αποτελεσματικότερο τρόπο για να προβάλλει κανεί την Ευρώπη. Θα υπάρχει κοινή σημαία και θα είμαστε πολύ πιο ορατοί από ό,τι είμαστε σήμερα. Στην περίπτωση τη ΕΤΗΣ εκεί ήμασταν πιο ορατοί. Η Χίλη είναι διαφορετική ιστορία. Ε, βλέπει κανείς τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, τα σύμβολα του Ερυθρού Σταυρού. Σε τέσσερα σημεία είδα το σύμβολο της Ευρώπης, τον πληρωνό με, τις, με τα στεράκια. Ε, το είδα σε ένα καταβλισμό, ε, σε μία δεξαμενή νερού, όχι σε δύο καταβλισμούς ε, σε μία δεξαμενή νερού και σε μία εγκατάσταση που είχαν εκεί ε, κουζίνας. Αυτά. Απλά για να τελειώσω αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, η δική μου η πρόθεση είναι να συνεργαστούμε στενά και με την κυρία Μάστρομ, γιατί αυτή ασχολείται με τη ρήτρα αλληλεγγύης και υπάρχει και εκεί ένα θέμα να έχουμε μια πολύ πρακτική προσέγγιση. Εμείς ελπίζουμε στις 22 Μαρτίου να βάλουμε σε πλαίσιο τη συζήτηση τις εναλλακτικές λύσεις και να πάρουμε εντολή από το Συμβούλιο Υπουργών έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε λεπτομερέστερη παρουσίαση ε, των σχεδίων. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ισπανική Προεδρία. Θέλουμε κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία να προχωρήσει η συζήτηση και επίση θα ήθελα να δράξω και την Ισπανική Προεδρία, Προεδρία να την ευχαριστήσω για το ότι ήταν ε, ιδιαίτερα ένθερμη σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά τώρα το κατά πόσον η κυβέρνηση να είναι σε θέση ή όχι να αποτελεί ισότιμο εταίρο όσον αφορά την ανοικοδόμηση της χώρας. Στην αρχή δεν είχαμε πολλές δυνατότητες και πράγματι χτυπήθηκαν πολύ σκληρά από τον σεισμό γιατί ε, τα κτίρια, τα περισσότερα κυβερνητικά κριτήρια έψαν πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων, σχεδόν κυριολεκτικά. Ε, και αυτό έγινε πριν από τι 5 η ώρα, ότι οι άνθρωποι είναι ακόμα στη δουλειά. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά για τη δημόσια διοίκηση, αλλά θέλω να πω το εξή. Στην IT είδαμε κάτι που εγώ δεν το ήξερα και με άγγιξε πάρα πολύ. Είδα ανθρώπους, πολίτες, οι οποίοι αυτοπροσδιορίστηκαν ηγέτες, αρχηγοί, ε, σε επίπεδο κοινότητας, σε μικρούς καταβλισμούς, όπου οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, πήγανε από κοινού στους καταβλισμούς από αυτού και ένας εξ αυτών αναλάμβανε να ε, μοιράσει δίκαια τα τρόφιμα, ε, τις δουλειές. Υπάρχει λοιπόν μια δικαιοσύνη στον επιμερισμό της εργασίας. Πρέπει να δεχθούμε ότι σε εθνικό επίπεδο υπολείπονται βέβαια πάρα πολλά, καλά, πάρα και είναι πολύ σημαντικό ε, οι ε, οργανισμοί, οι θεσμοί να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Αλλά το θέμα δεν είναι να δούμε τι κάνουν οι εθνικοί φορείς, να δούμε προς τα κάτω τι ακριβώς μπορεί να γίνει, να κινητοποιηθούν οι ηγετικέ δυνατότητες που υπάρχουν, κάτι που εμάς μας εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το θέμα είναι η κυβέρνηση μπορεί να προσφέρει σήμερα τη λήψη των αποφάσεων. Αυτό είναι δύσκολο. Πάντως θέλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα από ε, τον Πρωθυπουργό, ε, πάρα πολύ λειτουργικός, με πρακτικό πνεύμα, ε, ε στην ε, ε, αλληλεγγύη και την επικοινωνία. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και από τη Δομινικανή Δημοκρατία, γιατί ξέρετε πολύ καλά οι σχέσει μεταξύ των δύο κρατών κατά παρελθόν υπήρξαν προβληματικέ. Τώρα όμω ο σεισμό ένωσε τι χώρε αυτέ και υπάρχει ε, ουσιαστική επιθυμία στη Δομινικανή Δημοκρατία να βοηθήσουν. Και υπάρχει το θέμα της γλώσσας βέβαια σχετικά με τις δύο αυτές χώρες. Τέλος, Είχαμε μία συζήτηση σύντομη με τον νέο πρόεδρο και μου είπε «Φοβήθηκες» με ρώτησε. Του είπα δεν μπορώ να φοβάμαι. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τη διαχείριση κρίσεων. Δεν επιτρέπεται να φοβάμαι. Πάντως, οι άνθρωποι στη Χιλή έζησαν αυτόν τον τραγικό σεισμό του 8,8 και αυτοί ε, μας έκδοσαν θάρρος, γιατί αυτοί δεν φοβήθηκαν. Αυτό λοιπόν ήταν μια πραγματική ανθρώπινη επίδειξη θάρρους. Έξι ακόμη συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε σύντομοι στα ερωτήματά σας. Κύριε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να, να επανέλθω σε αυτό που έθεσε ο κύριος Μαρτίνες ε, για τους πυροσβέστες. Μας έκανε εντύπωση που δεν χρειάστηκε τα διασωστικά μας ε, ε, συνεργεία η χιλή. Πολλοί διασώστες έφτασαν στην Αϊτή όμως και φάνηκε ότι τελικά δεν τους χρειαζόταν η χώρα γιατί δεν, υπήρχε μεταφορέ, δεν υπήρχαν μεταφορές, δεν, υπήρχαν, ε, δεν υπήρχε σωστή επιμελητεία και δεν υπήρχε και μεταφορά επίσης ε, ξανά στο αεροδρόμιο. Δεν έφτασαν λοιπόν μέχρι τους ανθρώπους ε, που τους χρειάζονταν, τους ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε τρόφιμα και έπρεπε τελικά οι άνθρωποι να βοηθήσουν τους διασώστες που είχαν έρθει από άλλα μέρη του κόσμου ή από την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν περίεργο κάπως. Δεν είναι δυνατόν να παρέχουμε τέτοιου είδους βοήθεια κατά παραγγελία και μετά να περηφανευόμαστε ότι πω πω τι καλά που τα καταφέραμε και να ε, συγχαίρουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας. Ε, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε σωστά, δεν έχει κανένα νόημα και είναι και άχρηστο σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρετού έχει το λόγο. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, doamnă comisar. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, για την παρουσίασή σας και μια και μιλάμε, γιατί, ε, και αν μιλάμε, μια και μιλάμε για την ανθρωπιστική βοήθεια με την ευρύτερη έννοια, θα ήθελα να υποφεληθώ για να σας ρωτήσω η πτυχή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ποιο βαθμό ε, είναι παρούσα στην επίσκεψη που έκανε στη Μέση Ανατολή η κυρία Άστον. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο το θέμα που συζητούμε δεν είναι μόνο οι σεισμοί. Υπάρχουν ε, καταστάσεις που τις αντιμετωπίζουμε χρόνια. Στην Παλαιστίνη, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 500 εκατομμύρια σε προγράμματα εκπαίδευσης, ε, σε προγράμματα που προορίζονται για τις ευάλωτες οικογένειες, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο φτάνει στον πληθυσμό ε, η βοήθεια αυτή. Γιατί αν έχω καταλάβει καλά, μέσω της κυβέρνησης ε, πηγαίνει η βοήθεια, αλλά από τότε που η Χαμάς ε, έχει αναλάβει, ε, έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια της, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούμε να επαληθεύουμε την αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσίμερ έχει το λόγο. <clears throat> Mm, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω, καταρχάς, ότι πραγματικά δείξατε ιδιαίτερη αποφασιστικότητα στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου σας. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι μας δείξατε, προσπαθήσατε να μας δείξετε και είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με κάτι τέτοιο και δείξατε ότι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής ε, λειτουργήσε τελικά ή εν πάση περιπτώσει έγιναν πολλέ προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως να μου πείτε το εξή. Στην πρώτη σας αυτή η εμπειρία συνεργασίας υπήρξαν συμπεράσματα για τη μεταγενέστερη χρήση πόρων όσον αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων, για παράδειγμα, στους διάφορους τομείς. Και επίσης, Υπάρχει για το θέμα της βοήθειας για την ανοικοδόμηση. Η μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια στη βοήθεια για την ανοικοδόμηση ενδεχομένως να πάρει λίγο χρόνο. Και επίσης δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς που είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο. και δεδομένου ότι έχουμε και τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της IT... θα ήθελα να μάθω ποια θα είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διάσκεψη αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε μετά το μεγάλο τσουνάμι Μήπως σκεφτήκαμε να υπάρξει ένα μέσο διευκόλυνσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πώς το μέσο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Εν ολίγης, ποια είναι τα μέσα τα οποία θα είχε στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εμπειρία αυτή που είχαμε με το τσουνάμι για παράδειγμα είχαμε δυσκολίες γιατί το, τα κονδύλια δεν ήταν επαρκή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να το οργανώσουμε καλύτερα αυτό για το μέλλον. Θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε και για την προστασία των ε, φυσικών ε, καταστροφών. Όμως, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς από τη δική σας εμπειρία εφαρμόζετε τα μέτρα πρόληψης. Μιλήσατε βέβαια και για μέτρα εκτάκτου ανάγκης, αλλά τα μέτρα της πρόληψης τι θέση έχουν στην όλη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προβλέψουμε τέτοιου είδους θεομηνίες στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα έχω την εντύπωση ότι απαντήσατε στο ερώτημα που σας είχα θέσει στην πρώτη μας συνάντηση με την εξαγγελία του ανθρωπιστικού δόγματος, του ευρωπαϊκού ανθρωπιστικού δόγματος όπως το έχετε θέσει και χαίρομαι πάρα πολύ. Ήθελα να σας πω ότι στην τελευταία σύνοδο των Ασιατικών Κοινοβουλίων που είχα λάβει μέρος αποφασίστηκε η δημιουργία ενός task force το οποίο θα εδρεύει σε κάποια κέρια σημεία της Ασιατικής Υπήρου και είναι αυτό για το οποίο σας είχα μιλήσει την πρώτη φορά που να μπορεί να αντιδρά άμεσα εκείνο που έχει σημασία στους σεισμούς και βλέπω ότι το κλίμα έχει μεταστραφεί ανάμεσα στους συναδέλφους γιατί στις προηγούμενες συζητήσεις υπήρχε μια απογοήτευση για την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει άμεσα για την κρίση που ε, υπήρξε στη Χιλή, στην Αϊτή και όπου αλλού υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει η δύναμη εκείνη που να μπορεί να παρέμβει το πρώτο 24ωρο, το πρώτο 48ωρο. Από εκεί και πέρα εξαρτάται πιο πολύ από τις βασικές υποδομές της κάθε χώρας, όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει τη διαφορά ανάμεσα στην ΑΙΤΗ και στην Χιλή. Πριν από 13 χρόνια εργαζόμουν στην ΑΙΤΗ και είχα δηλώσει επιστρέφοντας ότι είναι ζήτημα χρόνου το πότε θα επισυμβεί αυτή η καταστροφή είτε με τη μορφή σεισμού είτε με τη μορφή των ε, κατολιστήσεων που ξέρετε πώς είναι διαμορφωμένο το έδαφος της χώρας αυτής και την καταστροφή των δασών. Συνεπώς, εκείνο που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε τις βασικές υποδομές σε κάθε χώρα Ενισχύοντα την δημοκρατία. Μην ξεχνάτε του Ντιβαλιέ που, είχαν αυτοί, που είχε η IT, μην ξεχνάτε την κακή διοίκηση του Αριστίτ και όλα όσα ακολούθησαν. Καθώ επίση και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων με τρόφιμα, φάρμακα και ή δυνατόν με πλωτά νοσοκομεία και πτυτικά μέσα, ιτάμενα ε, ε, νοσοκομεία. Τώρα, δύο παρατηρήσει όσον αφορά την Παλαιστίνη, την ξεχάσατε από την αρχική σας τοποθέτηση ενώ έχουμε μια μόνιμη ανθρωπιστική κρίση για την οποία δεν ευθύνεται καθόλου ο λαός της Παλαιστίνης. Και για να μπορούμε να ελέγχουμε τη Χαμάς ή την όποια Χαμάς ή την όποια Φάνταχ για την διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι φτάνει στην χώρα η ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ αμφιβάλλω αν περνάει την χώρα με το εμπάρκο που επιβάλλει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, ειδικά στην Λωρίδα της Γάζας. Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες από τις 27 χώρες δεν είχαν λάβει μέρος στην προσπάθεια για την ανακούφιση της χιλής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, με συγχωρείτε της ΑΕΤΙΣ. Είχατε πει 25 από τα 27 κράτη. Ποια ήταν τα δύο που δεν έλαβαν μέρος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργίευα, εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα είστε μια πολύ αφοσιωμένη επίτροπος και ότι θα επενδύσετε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει από τα προηγούμενα καθήκοντά σας και τα συναισθήματά σας στα σημερινά σας καθήκοντα, αλλά τώρα Εδώ μιλάμε πιο συγκεκριμένα για δύο καταστροφές που έγιναν ταυτόχρονα. Θα μπορούσαν να είναι και έξι και δεν θα μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε με τους ίδιους πόρους ε, και με το ίδιο επίπεδο οργάνωσης, ε, ούτε να ε, είμαστε στην ίδια κατάσταση παγκόσμιας ετοιμότητας, να συνεργαστούμε και να ελέγξουμε τέτοιες κρίσεις. Επίσης, είναι προφανές από το πόσα είπατε ότι αναμένουμε να συμβαίνουν ε, συχνά καταστροφές. Πριν ε, ένα-δύο χρόνια κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί τέτοιες καταστροφές όπως το τσουνάμι. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα χτυπήσει ένα σεισμός αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένα μέρη του κόσμου όπου οι καταστροφές είναι μόνιμες και μάλιστα είναι και πολύ χειρότερες καταστροφές από αυτές της χιλής της Αιτής. Σε σχέση με όσα είπαν ε, οι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω ότι μερικές φορές έχω το, την εντύπωση ότι μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, να βοηθήσουμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά αυτό οδηγεί στο να θέτουμε πάρα πολύ ψηλούς στόχους ε, ενίοτε. Με την ανθρωπιστική βοήθεια ε, δεν ε, είναι εύκολο να φέρουμε τον παράδεισο στη γη για τις χώρες που είναι υποανάπτυκτες, όπου υπάρχουν ε, τέτοιου είδου προβλήματα. Στην περίπτωση τη IT, να ρωτήσουμε ε, και τι έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείες τόσα χρόνια προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της ΑΕΤ. Έτσι λοιπόν, ενδιαφέρονται κάποιοι περισσότερο ίσως για τα χρήματα και για τις θυσίε που θα κάνουν προκειμένου να βοηθήσουν. Θα προσπαθήσω τώρα να είμαι πιο συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι χρειάζεται στενή συνεργασία παγκοσμίω και πρέπει να προβούμε σε ένα συντονισμό για το ποιος θα έχει την ηγετική θέση Νομίζω ότι και η διαχείριση των κρίσεων θα πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί νομίζω ότι αν γίνει μια κρίση στην Ασία, η Ιαπωνία θα έχει τον ηγετικό ρόλο για το συντονισμό. Αν γίνει στην Αμερική, πιθανότατα οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έχουν αυτόν τον ηγετικό ρόλο και εμεί θα έχουμε ηγετικό ρόλο στο δικό μα ε, τμήμα του κόσμου και πιθανότατα ακόμη και όλοι μαζί δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Αφρική. Δεν θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την Αφρική. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτή τη μόνιμη κρίση στην Παλαιστίνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πολιτικούς ε, λόγους έχουμε ανθρωπιστική καταστροφή. Αντίστοιχη με ε, ένα σεισμό 9 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Αν δηλαδή μιλάμε εδώ για το πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις ανθρωπογενείς καταστροφές. Και είναι και αποτέλεσμα μάλιστα κακής άσκησης πολιτικής. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ ευχαριστώ που μας ε, δώσατε τόσο ε, χρήσιμες πληροφορίες και δείχνετε και αυτή την ιδιαίτερη δέσμευση στο έργο σας και προσήλωση. Ευχαριστώ και τον κύριο Μαρτίνες ε, που εξήγησε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην IT και τη χιλή. Αυτό δεν θίγεται συχνά. Όταν γίνεται λόγος για την IT, πολλοί υπογραμμίζουν το θέμα της αγκληματικότητας και γνωρίζουμε ότι η IT αρκετό καιρό έχει πρόβλημα εγκληματικότητας. Γνωρίζουμε επίσης ότι ποια είναι τα αίτια. Τώρα πρόκειται για παιδιά τα οποία πολλούνται, έχουμε να κάνουμε με ομήρους, με εκβιασμούς, διακυβεύονται οι ανθρώπινες αξίες, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια η οποία καταπατάται με το χειρότερο τρόπο. Αυτό είναι πολύ χειρότερο από υλικέ ζημιές, όσο και αν είναι αυτές σοβαρές. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο το εξής. Εσείς σε ποιο βαθμό προβάλλετε τις ανθρώπινες αξίες που όπως σας είπα αποδοπατούνται με το χειρότερο τρόπο. Είναι δυνατόν ε, μεγαλύτερη βοήθεια να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εγκληματικότητα αν η τελευταία δεν αντιμετωπιστεί. Πολλοί αναφέρονται σε συμμορίες εγκληματιών που ε, εμφανίστηκαν, ε, συστάθηκαν εκ του συστάδιν. Ε, ίσως λοιπόν μπορεί η κυρία Επίτροπος να τοποθετηθεί από αυτού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ίσως επαναλαμβάνουμε, αλλά είπα στην Επιτροπή και τα προηγούμενα χρόνια για την ανθρωπιστική βοήθεια ότι κατ' ουσία κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ε, επανακαλύπτουμε τον τροχό. Είτε πρόκειται για το παλιροϊκό κύμα, είτε ε, για το σεισμό. Είπα λοιπόν προηγουμένως ότι ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδό μας προετοιμασίας. Αν χρησιμοποιήσουμε το ναυτικό μας και κυρίως ε, τα αεροπλανοφόρα μας, ε, διότι υπάρχουν 12 περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κατά την περίοδο μιας κρίσης πρέπει να υπάρχει μεγάλη ετοιμότητα. Το μόνο που μπορεί να απομακρύνει αυτά τα μπετόν που πέφτουν και πάνω στους ανθρώπους είναι τα ελικόπτερα. Τα αεροπλανοφόρα εξάλλου έχουν και συστήματα παροχής ύδατος και αφαλάτωσης τα αεροπλανοφόρα και τα σκάφη έχουν εξάλλου ε, και γιατρούς ε, επιτόπου, ε, αδελφές νοσοκόμες. Εάν λοιπόν εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας στην ανθρωπιστική βοήθεια ή όποτε το κάνουμε, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα. Μπορείτε λοιπόν να δείτε ότι ένα ισπανικό αεροπλανοφόρο είναι στον Α ωκεανό, ένα άλλο στο Β ωκεανό και γυρνάνε τον κόσμο. Γυρίζοντας λοιπόν τον κόσμο πρέπει ε, να υπάρχει εκπαίδευση σε ανθρωπιστική βοήθεια στην περίπτωση που συμβεί κάτι. Ας πούμε στη Μοζαμβίκη όπου εκεί έχουμε φοβερές ε, ε πλημμύρες ε, και άνθρωποι ζουν πάνω στις κορυφές των σπιτιών και των δέντρων. Μπορούν να απομακρυνθούν λοιπόν μόνο με ελικόπτερα. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα και ειδική προετοιμασία για τη χρήση αυτών των ελικοπτέρων. Η πρόεδρος δεν χρησιμοποιεί μικρόφωνο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος θα αναλάβει την ηγεσία, πώς θα οργανώσουμε την ανοικοδόμηση της ΑΕΤ, ποιος θα είναι ο ρόλος του ΙΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Παγκοσμίας Τράπεζας. Έχουν συζητηθεί τα θέματα αυτά και μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά. Και έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε, για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. I will actually start from uh, the... Να ξεκινήσω από τα θέματα που έθεξε ο κ. Κασμάρεκ. Είπε ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμός, καλύτερο συντονισμός. Στην περίπτωση της ΑΕΤΙΣ πρέπει να είμαστε λιγότερο αυστηροί, γιατί κοιτάξτε, όλα κατέρευσαν. Εμείς ε, χάσαμε όλους τους ε, ε, αναπληρωτές εκπροσώπους μας ε, της Κομισιόν, χάσαμε περίπου 200 άτομα, ε, κενώθηκαν τα κτίρια μας, πήγαν όσοι επέζησαν στο Μαϊάμι. Έτσι λοιπόν υπήρχε έλλειψη οργάνωσης και για αυτού του λόγους, αλλά φυσικά δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία για το ότι οι σημερινές μας ικανότητες ε, συντονισμού είναι τόσο περιορισμένες. Ε, προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις ε, στους αρμοδίους, αλλά δεν έχουμε τα μέσα προκειμένου να διαχειριστούμε την κρίση με έναν τρόπο που να είναι πιο αποτελεσματικός όλοι όσοι μίλησαν για συντονισμό τα έδειξαν τα θέματα αυτά και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα. Και να επανέλθω στο ΣΥΠΟ κ. Μπέρμαν, γιατί και άλλοι ομιλητές αναφερθήκαν στις ζητήματα αυτά, ότι η πιθανότητα θα πρέπει να σκεφτούμε μια παγκόσμια απάντηση και μήπως κάποιες χώρες πρέπει να αναλαμβάνουν ηγεσία ναι, ε, έχετε δίκιο όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, όχι για ενόπλες συγκρούσεις, όπου η συμμετοχή του στρατού στην ανθρωπιστική δράση πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά όταν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, Σίγουρα η ΑΕΤ θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση αν ε, δεν ε, υπήρχε ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων ε, με τους κατάλληλους εξοπλισμούς, τους μηχανισμούς παροχής ύδατος κτλ. Πρέπει λοιπόν στη δράση αυτή να προβαίνουμε αρκετά γρήγορα γιατί ε, πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας του κόστους της παρέμβασης. Ε, κάποιοι σήμερα οι οποίοι δεν είναι υπέρ της παρέμβασης, ανησυχούν για την αύξηση του κόστους. Όμως εγώ είμαι πεπισμένη ότι αν έχουμε μία παγκόσμια προετοιμασία, τότε θα γλιτώσουμε και πόρους. Όμω, θέλω να είμαι ειλικρινή εδώ, θα αντιμετωπίσουμε την εξή πραγματικότητα. Οι Χώρε που έχουν ε, ε, πολλά μέσα μπορεί να φοβηθούν ότι ε, θα του ασκηθεί πίεση να αναλάβουν μεγαλύτερο άχθος από τις χώρες που έχουν λιγότερα μέσα. Και αυτό το θέμα μπορούμε να το, να το αντιμετωπίσουμε μόνο αν ε, υιοθετήσουμε ε, ισότιμους όρους για την κατανομή του άχθους και προσπαθήσουμε ε, από αυτή τη συζήτηση να προκύψει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Κάποιοι ανέφεραν τη Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη. Και συγγνώμη, ανέφερα τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν έδωσε έμφαση σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα τώρα ε, που έχουν περάσει μέρες ε, μετά από την έκρηξη βίας ε, στην περιοχή. Η κυρία Άστον θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και κυρίως ε, θα εξετάσει το θέμα της πρόσβασης για τους ανθρώπους που εργάζονται στην ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό όπως με τη Διεθνή Επιτροπή του Διεθνού Σταυρού, του Ερυθρού Σταυρού ε, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε συντενισμό μεταξύ κρατών μελών, κομισιών και ε, όσων ε, έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Είναι αλήθεια ότι αυτό που έγινε κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα της ανάληψης θητείας ήταν το εξή. Πράγματι, ασχοληθήκαμε περισσότερο με αυτές τις δύο μεγάλες καταστροφές κυριαρχούσαν αυτές, αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε μέρη όπου οι σειράξει οδηγούν στο να υποφέρουν οι λαοί. Και φυσικά το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον και φυσικά θα λογοδοτήσουμε, θα σας αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την ε, ε, ανάληψη δράσης όταν συμβαίνουν οι καταστροφές έναντι της ετοιμότητας της διαχείρισης των καταστροφών. Αν δούμε τις δύο καταστροφές, προκύπτουν τα ακόλουθα. Η Χιλή εφάρμοσε για χρόνια και χρόνια προγράμματα αναδάσωσης και ε, μπορούσαμε να δούμε πόσα πολλά πράγματα είχαν γίνει για την αναδάσωση των λόφων. Και φυσικά αυτό έγινε σε αντίθεση με την IT όπου η ε, αποψήλωση οδηγεί στη διάβρωση και όπως καταλαβαίνετε η διάβρωση οδηγεί σε καθολιστήσεις. Αν έχουμε μια συστημική προσέγγιση, τότε θα πρέπει να διερευνηθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που αυξάνουν τις αντοχές μιας χώρας στην στις φυσικές καταστροφές και με την αλλαγή του κλίματος ε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη αστίαση ε, στους τομείς αυτούς. Από όλου όσου ασχολούνται με τα αναπτυσσιακά. Τώρα, για τον Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, θα πρέπει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσα ακόμη να επισκεφτώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σκοπεύω να το κάνω ε, με ένα μήνυμα από τη Χιλή, γιατί η Χιλή μόλις ε, έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ενδιαφέρεται ε, στο να λάβει πόρους για τη δημιουργία θέσεων εργασία και για τη λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και πραγματικά θέλω να δω τι μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να το τους επισκεφτώ. Αλλά να σας πω ότι πρέπει να διερευνούμε, να βλέπουμε ό,τι κάνουμε από τη σκοπιά της αύξησης των αντοχών ε, μιας χώρας ε, στις ε, κλιματικές αλλαγές, του σεισμούς, σε οποιαδήποτε μορφή καταστροφής. Γιατί ένα δολάριο ή ένα ευρώ ή οτιδήποτε αν επενδύσουμε χρήματα στην ετοιμότητα, ουσιαστικά αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από τις επενδύσεις. Για το θέμα των υποδομών και την εταιρική σχέση με τις ασιατικές χώρες στον τομέα αυτό. Ένας από τους στόχους, και μπορώ να το δω αυτό από το παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής, ότι έχει ιδιαίτερο νόημα, γιατί το τμήμα του χαρτοφυλακίου μου που αναφέρεται στη διεθνή συνεργασία είναι να επεκτείνει τη συνεργασία, να διευρύνει τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Και φυσικά αυτή η ετοιμότητα έναντι των φυσικών καταστροφών ε, είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα. Να επιβεβαιωθώ ότι μπορώ να μεταβώ τώρα στην τελευταία ερώτηση. Συγγνώμη, ξέχασα την τελευταία ερώτηση της Πρόεδρου. Ναι, με συγχωρείτε. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έχουν θεσπιστεί 12 κλάστερς. Και μετά από κάποιες, ε, κάποια προβλήματα στην έναρξη τώρα υπάρχει ένας καλός συντονισμός ε, για το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας σε 12 τομείς. Εμείς ε, έχουμε τέσσερις τέτοιες ομαδοποιήσεις. Υπάρχει τώρα συντονισμός και τελικά ουσιαστικά παραμένουμε σε ένα πυρήνα των πλέον ενεργών συμμετεχόντων αρχικά μια τέτοια ομαδοποίηση είχε πάνω από 250 συμμετέχοντες. Φυσικά δεν μπορούσε να γίνει διαχείριση, όμως ε, υπήρχαν συντονιστικέ συναντήσεις στην ΑΕΤ και μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όταν ε, όμως ε, μιλάμε για μια μεγάλη προσπαθία νοικοδόμησης, να σας πω ότι έλαβα feedback από κάποιες αναπτυξιακές τράπεζες, την Αμερικανική Τράπεζα από τον ΟΗΕ και από την Inter-American Development Bank. Ε, όλοι αυτοί οι οργανισμοί ε, θα κάνουν μία μελέτη αντικτύπου για την ανάπτυξη και συστήνουν μία κοινή ομάδα και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τις ικανότητες τη κυβέρνηση Η κυβέρνηση δέχεται ότι πρέπει να συνεργαστεί με άλλου φορεί και η μελέτη αυτή θα παρουσιαστεί στις 31 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, αλλά νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμη και νωρίτερα. Είναι θα είναι διαθέσιμη συνάντηση στον Άγιο Δομηνικό που θα λάβει χώρα αύριο. Και Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και στη συνδιάσκεψη της Νέας Υόρκης. Στη μελέτη αυτή προσπάθησαν να εντοπίσουν προτεραιότητες και να προβούν σε κατανομή ευθυνών. Πολλές ε, φορές ε, ξέρετε ότι ε, στον τομέα της ανάπτυξης φαίνεται σαν να παίζουμε ποδόσφαιρο, δηλαδή εκεί που είναι η μπάλα όλοι είναι μαζεμένοι γύρω-γύρω. Όμως να πω και κάτι ακόμη για την IT. Νομίζω ότι η βία και το έγκλημα αποτελούν πρόβλημα, αλλά η καταστροφή σε πάρα πολλές περιοχές ε, οδήγησε στη σύσφυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Εμείς στην Κομισιόν ε, θέτουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα προστασίας των παιδιών, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα Είδα ε, διάφορες περιοχές ε, στην ΑΕΤ, κάποια μέρη όπου εγώ δεν θα έβγαινα έξω στο σκοτάδι και κάποια μέρη όπου κάποιος ε, αισθανόταν ε, τη ζεστασιά των ανθρώπων. Δεν έμεινα πάρα πολύ για να σχηματίσω οριστική άποψη, αλλά μπορώ να σας πω ότι όταν ε, υπάρχουν άνθρωποι που οποίοι λαμβάνουν δράση ήταν ε, πολύ καλύτερο το περιβάλλον ενώ σε άλλα σημεία πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνουν βιασμοί και να πάγονται παιδιά. Το πώς, πώς απαντάμε τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθούν σωστά οι δυνάμεις ασφαλείας και φυσικά ο ΙΕ έχει την ευθύνη και την ηγετική θέση. Ο ΙΕ προσπαθεί να διανύμει να αναπτύξει ε, τις δυνάμεις ε, προστασίας ε, με έναν τρόπο αποτελεσματικό και αναλογικό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. θα ήθελα και εγώ να πω κάτι που αφορά στην απάντηση που πήρα για την οργάνωση. Κοιτάξτε, από τη δική μου εμπειρία, από τη Νορβηγία, γνωρίζω ότι τα Ηνωμένα Έθνη ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο να γίνεται κάτι. Όχι δε, όμως δεν ισχύει το ίδιο για την Παγκόσμια Τράπεζα, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρω ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων προτιμάει ε, την Παγκόσμια Τράπεζα από τα Ηνωμένα Έθνη και θα σκίσουν πίεση και στις δύο χώρες που πέσαν σεισμό έτσι ώστε ε, εκεί να καταφύγουν για το μοντέλο νοικοδόμηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ως εκ τούτου η δική μας η Επιτροπή ε, πρέπει να επαγρυπνεί όσον αφορά ε, αυτό το θέμα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι για ερωτήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που πήρατε. Ε, πάντα είναι ιδιαίτερα λεπτό το θέμα το να επικρίνει κανείς άλλους διεθνείς οργανισμούς. Πιστεύετε ότι είναι σοφό το κεφάλαιο της IT ε, και του Port Brown να συγκεντρωθούν στο ίδιο ακριβώ σημείο όπου υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα και υπάρχει και ουσιαστικός κίνδυνος να επαναληφθεί αυτός ο καταστροφικός ε, ε, σεισμός. Εγώ θα έλεγα να μεταφερθούν οι πληθυσμοί σε ένα ασφαλέστερο σημείο. Κοιτάξτε, για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όσους μετακινήθηκαν από το Πορτοπράνς να παραμείνουν εκεί που μετακινήθηκαν. Αυτό το όλο θέμα της ανοικοδόμησης της IT της ε, αν πρόκειται να γίνει όπως ήταν και παλιά, ε, γιατί να χρησιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι πόροι. Εγώ δεν ε, ξέρω αρκετά στοιχεία για να μπορώ να σας πω ε, πόσο ασφαλή ή ασφαλέστερα είναι όλα τα σημεία του Πόρτο Πράνς. Όμως όταν πετάξαμε πάνω από την πόλη είδα περιοχές που ήταν απόλυτα κατεστραμμένες, ερήπια και άλλες που δεν ήταν τόσο κατεστραμμένες. Άρα δηλαδή βλέπει κανείς ότι πρόκειται για μια, ε, ένα πρανές όπου κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Και αυτό ε, είναι πάρα πολύ ε, κρίσιμο. Εγώ πιστεύω ότι ε, για να υπάρξει ανοικοδόμηση πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σε σχολείο. Γιατί να μην έχουμε στόχο την επόμενη χρονιά τα παιδιά να έχουν πάει όλα σε σχολείο και τα σχολεία αυτά να είναι ασφαλέστερα. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό ε, ρεύμα. Τώρα οι άνθρωποι υποφέρουν στην ΑΕΤ γιατί δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί λοιπόν σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια να μην ε, τοποθετηθούν ε, ηλιακοί συλλέκτες ή το θέμα της αποψήλωσης. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μερικές φορές, όταν οι αναπτυξιακοί φορείς ε, συνεργάζονται, τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Επιτροπή, ε, μπορούν να κάνουν θαυμάσια πράγματα. και αυτο μπορει να αντιμετωπιστει μερικες φορες οταν οι αναπτυξιακοι φορεις συνεργαζονται τα εθνη η παγκοσμια τραπεζα η επιτροπη μπορουν να κανουν θαυμασια πραγματα και το έχουμε δει αυτό μερικές φορές στο πλαίσιο της διαρκούς βιώσιμης και εφόρων ανάπτυξη ότι ε, μπορούν να επιτευχθούν πολύ σημαντικοί στόχοι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ΑΕΤ ε, θα είναι ένας ε, στόχος. Ο κύριος Φίσας, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. στην ε, ακρόασή σα για την ανέλεψη των καθηκόντων σα ω επίτροπε, είχα την ευκαιρία να σα ε, ρωτήσω για την κατάσταση των ε, κατοίκων τη Σαχάρα. Εσεί μα είχατε πει ότι δεν θα ξεχνούσατε αυτού του ξεχασμένου κατά κάποιο τρόπο από όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε αναλάβει κάποια δράση σχετικά με το ζήτημα αυτό, είχατε την ευκαιρία να ασχοληθείτε. Κοιτάξτε, η πολύ ειλικρινή απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κάνει ακόμη τίποτα. Όχι μόνο γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα έκτακτα γεγονότα, αλλά και γιατί, όπως ε, ενδεχομένως γνωρίζετε όλοι, ότι δεν είχα ομάδα, έπρεπε να διαμορφώσω μια ομάδα, να κάνω μια επιλογή ε, συνεργατών και να αντιμετωπίσω ζητήματα πολύ επίγοντα. Δεν το έχω ξεχάσει όμως, γι' αυτό ακριβώς είπα για ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και για τα οποία δεν έχουμε ακόμη παρουσιάσει ένα πολύ σαφές όραμα για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, θα επανέλθουμε. Εδώ είναι μάλιστα ο συνάδελφός μου ε, από την ομάδα μου υπεύθυνο ε, αναπληρωτής μου που τα σημειώνει όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ε, που ήρθατε να μοιραστείτε μαζί, μαζί μας την εμπειρία τις εμπειρίες σας και τις προτεραιότητάς σας και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα σας, σας ξαναέχουμε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, έχουμε μισή ώρα καθυστέρηση. Δεν ήθελα όμως να διακόψω τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα που είχαμε με την Επίτροπο. Θα περάσουμε τώρα στο δημοκρατικό έλεγχο των μηχανισμών ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα ακούσουμε τα συμπεράσματα των ομάδων εργασίας Α, Γ και Δ. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή, η Επιτροπή μας από την αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας έχει ε, ιδρύσει πέντε ομάδες ε, εργασίας μόνιμες για τον δημοκρατικό ε, έλεγχο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του άρθρου 88 του εσωτερικού μας κανονισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αναπτυξιακή συνεργασία. Πρόκειται για τα μέτρα επιτροπολογίας τα οποία μας υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν έγκριση των κρατών μελών στο πλαίσιο της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης. οι ομάδες αυτές ε, προβαίνουν σε έναν ε, διαρθρωμένο και μόνιμο κατά κανόνα διάλογο και πρέπει βέβαια σε ένα πρώτο επίπεδο να ακούσουμε τα μέτρα τα εκτελεστικά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, βέβαια υπό το φως των πολιτικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βέβαια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Κάτι άλλο το οποίο είναι πιο τεχνικό, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πρόκειται για τις αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Έχουμε ένα δικαίωμα εξέτασης, δημοκρατικού ελέγχου για όλα τα προγράμματα εκτελεστικών μέτρων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Διαχειριστική Επιτροπή για την εφαρμογή των διαφόρων μέσων. Σας υπενθυμίζω ότι οι διαχειριστικές αυτές επιτροπές αποτελούνται από εκπροσώπους των κρατών μιλών ε, και την Προεδρία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του δικαιώματο εξέταση, πρέπει εντό 30 ημερών μετά την έγκριση των κρατών μελών, στο πλαίσιο τη Διαχειριστική Επιτροπή, ε, να προτείνει ένα, να γνωμοδοτήσει επί του προτινόμενου μέτρου εμπροκειμένου στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης ε, και συνεργασίας και ανάπτυξης ε, στο πλαίσιο της, ε, του μέσου διευκόλυνσης για τα τρόφιμα. Υπάρχουν τρία πακέτα μέτρων στο πλαίσιο των στρατηγικών εγγράφων, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της μεσοπρόθεσης των εγγράφων της γεωγραφικής και, στρατηγική, και θεματικής στρατηγικής, όπως επίσης και ένα τέταρτο πακέτο των μέτρων που ιδρύει ένα μέσο για την ε, επιζητιστική βοήθεια. Οι ομάδες αυτές ε, παρουσίασαν ε, τα συμπεράσματά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την πρώτη. Η κυρία Θεοχάρους θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ε, συνεδρίασης της ε, Επιτροπής της ε, με την Επιτροπή της Μαρτίου. Έχετε το λόγο. Uh, well, dear colleagues, working group A. Ευχαριστώ. Η ομάδα Α συναντήθηκε στις 3 Μαρτίου για να συζητήσει το ενδεικτικό πρόγραμμα για την Κεντρική Ασία για το 2011-2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης συμμετείχε στη συνάντηση αυτή ένας συγκεκριμένος στόχος του Περιφερειακού Ενδικικού Προγράμματος για την Κεντρική Ασία ήταν να καταπολεμήσει τη διεθνή τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και την ε, διακίνηση όπλων ναρκωτικών ε, και την εμπορία ανθρώπων ε, και εφαρμόζοντας ε, συστήματα ε, για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Ε, εμείς για το πρόγραμμα 2011-2013 στοχεύουμε περισσότερο στην καταπολέμηση της, του οργανωμένου και της θερμοκρατίας μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα αυτό δεν συνάδει με τους κανονισμούς DCI για τους ακόλουθους λόγους. Όλα τα μέτρα καταρχήν που προτείνονται υπό το γεωγραφικό πρόγραμμα DCI θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που καταρτίστηκε από τον ε, ΟΣΑ. Δεύτερον, ε, το άρθρο 2 του DCI δηλώνει ότι τα μέτρα που καλύπτονται από τους κανονισμούς τα 17 του 2006 το μέσο για τη σταθερότητα και ε, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση δεν θα χρηματοδοτούνται από τον κανονισμό αυτό. Και τρίτον, το 2007 το ΔΕΚ στην υπόθεση C 405 ε, ε, αποφάσισε ότι παρόμοια μέτρα καταπολέμησης τρομοκρατίας που προτείνονται δυνάμει του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας από την Κομισιόν δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το μέσο αυτό στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Α, ζητήσαμε από την Κομισιόν να μας εξηγήσει για ποιο λόγο συμπεριέλαβε τα μέτρα αυτά στο ενδεικτικό πρόγραμμα. Η Κομισιόν παραδέχτηκε ότι τέτοια μέτρα δεν εμπίπτουν ε, για χρηματοδότηση υπό τον DCI και ε, προτέθηκαν για χρηματοδότηση υπό το μέσο Σταθερότητα η Κομισιόν υποσχέθηκε να αλλάξει το έγγραφο για την Κεντρική Ασία και να διαγράψει κάθε αναφορά στις δραστηριότητες καταπολέμησης τη Τρομοκρατία. Ζητούμε λοιπόν ε, τις για τα ακόλουθα συμπεράσματα. Καταρχήν, στο στάδιο αυτό τη διαδικασία διαβούλευση και βάσει των εγγράφων και των διαβεβαιώσεων που λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ομάδα Α δεν συστήνει στην Επιτροπή ανάπτυξη να υιοθετήσει το ψήφισμα δυνάμει του άρθρου του κανονισμού και Δεύτερον, η ομάδα εργασία μα προτείνει στην Επιτροπή Ανάπτυξη να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίε και αιτιολόγηση για το πιο γενικό θέμα τη συνεργασία στο τομέα τη ασφάλεια και την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων στην περιοχή τη Κεντρική Ασία και στι αναπτυσσόμενε χώρε εν γέννη και τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων. Και ε, φυσικά στις 21 ε, έχουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τις εκθέσεις για το λαό της Φιλιππίνες και τη Μογγολία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, να δει κανεί ο δημοκρατικός έλεγχος πόσο σημαντικό είναι για να γίνονται σεβαστοί οι κανόνε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενς, υπεύθυνο της ομάδας εργασίας ΔΕΛΤΑ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την γραμματεία και τους βοηθούς της ομάδας μας, όπως επίσης και τα μέλη της Επιτροπής. Ε, είχαμε μία συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, παρά το γεγονός ε, ότι η συμμετοχή δεν ήταν πάντοτε επιθυμητή. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε κατά την συνάντησή τους στις 3 Μαρτίου για τα εξή ζητήματα. Πρόκειται για την αναθεώρηση τη μεσοπρόθεσμη 2011-2013 για τη Βολιβία, αναθεώρηση μεθοπρόθεσμη των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων για την ίδια περίοδο για τη Βενεζουέλα και επίσης ε, η ίδια αναθεώρηση 2011-2013 για την ε, περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής. Κανένα από τα έγγραφα αυτά δεν φαίνεται να μπορεί να ε, μας δημιουργεί πρόβλημα. Εκτός από τα... Όσον αφορά τα εφαρμοστικά μέτρα, η ομάδα μας δεν διαφωνεί με τα σχέδια μέτρων, αλλά προτείνει μία σύσταση που ζητά την στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη ε, σοβαρά τις ε, προτάσεις μας. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες ιδιαιτερότητες ε, για το καθένα από τα έγγραφα αυτά και μετά θα σας αναφέρω τα συμπεράσματά μας σε σχέση με την στάση που προτείνουμε να ληφθεί για το σύνολο των εγγράφων αυτών. Πρώτον για τη Βολιβία. Η κυρία Κρετού ήταν η εισηγήτρια για το σχετικό έγγραφο της Βολιβίας. Και προτείνω να αρχίσουμε πρώτα οι κυρίε από το συγκεκριμένο έγγραφο, εκτό αν η κυρία Κρετού θέλει να το κάνει μόνη τη. Βέβαια δεν είναι εδώ. Οπότε νομίζω ότι θα το κάνω εγώ. Η Βολιβία είναι μία από τις στοχότερε χώρες της Λατινικής Αμερικανής και Αμερικής και αντιμετωπίζει οικονομικά, κοινωνικά ε, και πολιτικά προβλήματα για την περίοδο 2011 2013. Προτείνεται 115 εκατομμύρια ευρώ διόλο μελιτέο ποσό. Καταπολέμηση της φτώχειας, καταπολέμηση των ναρκωτικών και ε, αηφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ε, διαφωνεί με τα βασικά κριτήρια ανάλυσης που έχουμε. Πρόκειται για αναπτυξιακή βοήθεια στο πλαίσιο του ΩΣΑ και πρόκειται για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως επίσης και για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Υπήρξαν όμως και κάποιες ανησυχίες. ή εξής. Σε γενικές γραμμές ε, είναι δύσκολη η λεπτομερής αξιολόγηση γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς λεπτομέρειες ειδικότερα όσον αφορά τον εντοπισμό των ομάδων στόχο. Πρέπει να εδραιώσουμε την κρατική υποδομή να, υπάρξει, να υπάρξουν υποδομές και σε θεσμικό και σε νομοθετικό επίπεδο. Επίσης υπάρχουν και άμεση τρόποι, αμεσότεροι ενδεχομένως για την καταπολέμηση της φτώχειας που είναι η υποστήριξη στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά στη Βενεζουέλα τώρα, η κατάσταση της χώρας είναι πολύ ιδιαίτερη και σε μερικές περιπτώσεις ανησυχητική λόγω των ε, ε, της αναστάτωσης της οικονομικής, ε, κοινωνικής και πολιτικής ε, κατάστασης, ε, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ του Προέδρου Τσάβες και των ε, αντιπάλων του. 10 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν προβλέπονται, ένα τέταρτο του ε, φακέλου για την ε, περίοδο 2007 με 2013. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσό λοιπόν. Δύο βασικοί τομείς θα υποφεληθούν, ο εξυγχρονισμό και η αποκέντρωση από τη μία και από την άλλη οικονομική διαφοροποίηση οι δράσεις ε, που θα, οι δράσεις καλύπτονται από τον κατάλογο 4 του ΩΣΑ, που είναι ένα ζήτημα που θέτουμε συνεχώς. Καλύπτονται από τον κατάλογο λοιπόν αυτών ε, για τη δημόσια βοήθεια ε, για την ανάπτυξη και ελπίζουμε να μπορέσουμε περισσότερες λεπτομέρειες να έχουμε στο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί. Ε, υπάρχει επίσης, ε, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ε, για τα εξής ζητήματα. Δεδομένου του πλαισίου των περιορισμένων πόρων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ενώ στόχος, η χώρα στόχος είναι μία από τις πλουσιότερες της περιοχής, θα μπορούσαμε γενικά να αναρωτηθούμε εάν ε, αποτελεσματικά διαθέτονται οι πόροι αυτοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων, ε, των στόχων της χιλιετίας. Επίσης υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το εξής ασαφής χαρακτήρας των δικτών ε, για να μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε με δύσκολες, ε, με δύσκολες ε, πολιτικές αρχές στο πλαίσιο CAD... και οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Όσον αφορά λοιπόν τη συνεργασία, με τις χώρες δωρητές, ε, είναι σημαντικό να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι χώρες. Πρέπει να γίνει ένας πραγματικός διάλογος με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις τις τοπικές ε, και επίσης πρέπει να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τη δύσκολη κατάσταση της ε, Παρέμβαση τη κυβέρνηση, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης ένα θέμα που μένα με απασχολεί πάρα πολύ ένας ε, διάλογος ε, ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προγραμμάτων ε, μεταξύ της Βενεζουέλας και των φυσικών εταίρων της, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Αργεντινή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό, να υπάρξει δηλαδή συνεργασία μεταξύ της Βενεζουέλας και των τριών αυτών εταίρων της, θα μπορούσαν και εκείνες να είναι χώρες δωρητές ο ένας θα μπορούσε να είναι πάροχος υπηρεσιών ε, και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ε, μια ε, συνεργασία τριμερής υπ' αυτήν την έννοια. πέραν του κατά πόσο έχουν πλέον δικαίωμα σε αναπτυξιακή βοήθεια ή όχι, θα μπορούσαν μόνοι τους να συνεργαστούν μέσω αυτής της τριμερού συνεργασίας που προτείνουμε. Μία τρίτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, τρίτο σχόλιο, έχει να κάνει με την Λατινική Αμερική ολόκληρη δηλαδή την περιφέρεια αυτή. Είναι μια τεράστια περιφέρεια, ε, πάρα πολύ πλούσια Υπάρχει μια τάση περιφερειακής ολοκλήρωσης, όλες ε, οι χώρες ε, συμμετέχουν σε αυτή. Βέβαια υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, κρατών όσον αφορά τις δημοκρατικές αξίες και όσον αφορά τις οικονομίες αγοράς. Σε σχέση με το ΑΕΠ επίσης υπάρχουν διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη και επίσης υπάρχουν ρεκόρ κοινωνικής ανισότητας. 10% του πληθυσμού σε σχέση με 30 των στις βιομηχανοποιημένες χώρες έχουν 50% του πλούτου, πάνω από 200 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Ε, μιλάμε δηλαδή για τρομερές συνθήκες φτώχειας. 194 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ των δύο βασικών τομέων που έχει να κάνει με την περιφερειακή ολοκλήρωση, ε, τη συνεργασία, την αμοιβαία και την ανώτερη εκπαίδευση αν οι προγραμματισμένες δράσεις σε, αυτές, σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας εκπληρώσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΚΑΔ ε, για την δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, παρόλα αυτά η ομάδα εργασίας είχε επιφυλάξεις κατά πόσο οι προγραμματισμένες του τομέα δύο δράσεις, δηλαδή η αμοιβαία κατανόηση και η ανώτερη καλύτερη εκπαίδευση ε, υπάρχει στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Γι' αυτό η σύνδεση με την ε, ανάπτυξη ενώ υπάρχει δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσε να οδηγήσει στους ε, στόχους, στην επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών της χιλετίας. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν αυτό έχει να κάνει κυρίως ε, με το μέσο ενίσχυσης ε, στα πλαίσια της ανάπτυξης, περισσότερο δηλαδή έχει να κάνει με την αμοιβαία κατανόηση και επομένως θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί εκτός της αναπτυξιακής βοήθειας ε, η νέα προτεραιότητα της κλιματικής αλλαγής, που είναι κάτι νέο και για την περιφέρεια δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα και Όσον αφορά τα γενικά συμπεράσματα, η ομάδα εργασία, βάσει των εγγράφων που έχει λάβει, προτείνει στην Επιτροπή Ανάπτυξη να μην διαφωνήσει στο πλαίσιο τη διαδικασία επιτροπολογία ε, του άρθρου 5 και στο άρθρο, του άρθρου 88 του εσωτερικού μα κανονισμού, στα διάφορα εφαρμοστικά μέτρα τη αναθεώρηση μεθοπρόθεσμη ε, και της, του ενδεικτικού προγράμματο ε, που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βενεζουέλα ε, την Βολιβία και την Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι είναι ο πιο απλός τρόπος ε, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή Ανάπτυξης να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο DCI να υποβάλουν τις παρατηρήσεις αυτές στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των προγραμμάτων των ενδεικτικών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Τα μέλη που είναι παρόντα συμμερίζονται τις αναλύσεις ε, και τις απόψεις του κυρίου Γκέρες ε, για την ομάδα εργασίας ΔΕΛΤΑ. Μπορούμε λοιπόν να, να δεχτούμε ότι εγκρίνονται από την Επιτροπή. Ας ε, δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας C, ο κύριος Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η ομάδα ανέφερε την ευθύνη της απέντη που έχει στην ομάδα εργασίας και εμείς ασχολούμεθα με την Καράγουα, με την Κούβα σε αυτό το έγγραφο ε, περιφερειακής στρατηγικής για την ε, Κεντρική Αμερική, για τη Γουατεμάλα. Ασχολούμεθα επίσης ε, με το έγγραφο στρατηγικής που έχει ως θέμα τη μετανάστευση και το άσυλο. Και επίσης και για το Ελσαλβαντόρ, το Μεξικό, την Κοσταρίκα και τον Παναμά. Σήμερα το πρωί η ομάδα εργασίας αξιολόγησε και σχολίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης ε, με τους εκπροσώπους Εκτελεστικής Επιτροπής. Αναφέρθηκε επίσης ε, στα προσωρινά συμπεράσματα ε, και μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η περιφερειακή στρατηγική της Επιτροπής παραμένει αμετάβλητη. Η ενίσχυση του θεσμικού συστήματος προς όφελος της ενσωμάτωσης ε, της ολοκλήρωσης στην Κεντρική Αμερική, η ενίσχυση της διαδικασίας οικονομικής ολοκλήρωσης, ενίσχυση της ε, περιφερειακής ασφάλειας. Όσον αφορά κυρίως αυτό το τελευταίο θέμα, δηλαδή την περιφερειακή ασφάλεια, η ομάδα εργασίας είναι ιδιαίτερα ε, προβληματισμένη όσον αφορά τον περιορισμό της ένδυας, αλλά επίσης και την επίτευξη των στόχων της χιλιοετίας σχετικά με την ανάπτυξη. Το Κοινοβούλιο το 2007 επισήμανε ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτών των στόχων ε, δεν είχαν άμεση σχέση με τον κοινωνικό τομέα, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, και παρά την κρίση στα τρόφιμα και στην οικονομία που ολόκληρη η περιοχή αντιμετωπίζει από το 2008, κανένας από τους ε, πρωταρχικούς ε, στόχους ε, της, του εγγράφου για την περιφερειακή στρατηγική δεν συνδέεται, κανένας λοιπόν δεν συνδέεται με την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας πέρα από αυτό, ε, εξεργουμένη της Ονδούρας και εν μέρει και της Νικαράγος, όπου η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται ως προτεραιότητα, η περιγραφή των δράσεων του ε, στρατηγικού, εθνικού στρατηγικού εγγράφου δεν είναι άμεσα συνδεμένη με τον περιορισμό της φτώχειας και την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Όσον αφορά στο θέμα αυτό, η Επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι χορηγοί που ασχολούνται με το θέμα της υγείας και της ε, εκπαίδευσης. Η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, ένα πολύ, ένας πολύ ευρύς όρος που όπως πολύ καλά γνωρίζετε περιλαμβάνει θέματα που αρχίζουν από την περιφερειακή ανάπτυξη και φτάνουν μέχρι την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό πρόσφατα είχε θετικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι η πρωταρχική ε, τομείς ε, έχουν σχέση με το θέμα της συμβατότητας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης πέρα από τα προβλήματα που απαριθμεί στον τομέα αυτό και στο έγγραφο που εξετάστηκαν, αναφέρει ότι ε, αυτά είναι συμβατά και πρέπει να είναι συμβατά με τους ε, στόχους της ανάπτυξης. Όσον αφορά τις βασικές αλλαγές ε, μέσω πρόθεσμα, αυτό που παίζει ρόλο είναι η εφαρμογή των κονδυλίων του Ταμείου για επενδύσεις στη Λατινική Αμερική. Αυτό το Ταμείο θα λάβει πόρους από την Επιτροπή, μάλλον από το εργαλείο ανάπτυξης για να προαχθεί η ολοκλήρωση της ε, κοινή αγοράς στην Κεντρική Αμερική. Η δική μας λοιπόν η ομάδα ε, θεωρεί ε, ότι μπορεί να διαβεβαιώσει ότι τα κονδύλια αυτά θα διοχετευθούν κυρίως στον αγώνα κατά της ένδυας. Η ομάδα ανησυχεί για το ότι τουλάχιστον τρεις χώρες, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα και η Νικοράγωα, αυτές οι τρεις χώρες είχαν δυσκολίες στο να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια που διοχητεύτηκαν ε, για τον ισοσκελισμό του ε, προπολογισμού. Σε πολλές περιπτώσεις τα κονδύλια αυτά αντικαταστήθηκαν από ε, άλλα σχέδια που έχουν ως στόχο που δεν έχουν ως στόχο την ενίσχυση και τον ισοσκελισμό του προπολογισμού έτσι ώστε να προαχθεί ο πολιτικός διάλογος. Όσον αφορά τώρα τους διάφορους παράγοντες, η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι στην περίπτωση της ε, κοινωνίας των πολιτών οι διαβουλεύσεις θα έπρεπε να οργανωθούν αρκετά έγκαιρα με προειδοποίηση. Τα βασικά έγγραφα θα έπρεπε να έχουν διατεθεί στις ε, γλώσσες ε, των χωρών αυτών ή των περιοχών. Τα κριτήρια για προσκλήσεις θα έπρεπε να είναι σαφή, να είναι αρκετά εκτεταμένα τόσο όσο τον κατάλογο όσο και τις διαβουλεύσεις όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν κοινοποιηθεί. Εξάλλου η ομάδα εργασίας ανησυχεί διότι μόνο λίγα κοινοβούλια συμμετείχαν ε, σε αυτή την αναθεώρηση και τα βασικά αίτια αυτού είναι ότι υπήρξαν δυσκολίε στο να συμπεριληφθούν αυτοί οι θεσμοί και στο ότι δεν υπήρξε επαρκής διαρθρωμένος διάλογος ανάμεσα σε αυτές και ε, την Εκτελεστική Επιτροπή. Εξάλλου επισημαίνεται ότι η ανάλυση αλλά και οι συζητήσει που έλαβαν χώρα στα πλαίσια ενός διαρθρωμένου διαλόγου ε, θα έπρεπε να βασίζονται στη διαφάνεια και στην ανταλλαγή απόψεων. Έτσι λοιπόν εμεί εκφράζουμε την επιθυμία στο μέλλον η Επιτροπή και η ομάδα εργασίας για τη διαχείριση του εργαλείου σχετικά με τη συνεργασία και την ανάπτυξη, αυτοί να προσφέρουν ε, πιο επικαιροποιημένα και ε, πλήρη κείμενα. Οι συστάσεις λοιπόν προς την Επιτροπή Ανάπτυξης είναι σε αυτό το σημείο τις βάσεις διαβουλεύσεων και με βάση τα έγγραφα που έχουν, ε, έχουμε στα χέρια μας λέμε ότι δεν θα πρέπει να εκφράσουμε αντιρρήσει απέναντι σε αυτό το εθνικό ε, έγγραφο το Παναμά, Γουατεμάλα, Ονδούρας, Μεξικό, Κωνσταρίκα, ω ως ε, ε, ένα σημαντικό έγγραφο της Κεντρικής Αμερικής και τούτο στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας που προβλέπεται από το άρθρο 35 του καταστατικού και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ομάδα ζητά από την Επιτροπή Ανάπτυξη να ενημερώσει τα κράτη-μέλη και όλους του άλλου αρμόδιου και εμπλεκόμενους φορείς ε, το τι ακριβώς ε, έχει προκύψει από τις αναλύσεις λαμβάνοντας κυρίως υπόψη το τι είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη σχετικά με αυτό το εθνικό ε, και περιφερειακό έγγραφο. Τα μέλη συμφωνούν με την ανάλυση της ομάδας εργασίας ΣΥ. Μάλιστα, θετούμε λοιπόν τις συστάσεις αυτές. Το λόγο τώρα έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Κύριος Πένιντον, και αν μπορείτε σας παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Απλώς, ε, συντομία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη αυτών των διαφορών ομάδων εργασία ε, για την προσπάθεια που κατέβαλαν, ε, για την διεξαγωγή του διαλόγου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αλληλεπίδραση στο επίπεδο αυτό και να μας γνωστοποιείτε τις ανησυχίες σας. Εγώ συμμετείχα στις εργασίες της ομάδας Α. Ευχαριστώ την κυρία Θεοχάρους για τη σύνοψη. Η Κομισιόν δέχεται όλες τις παρατηρήσεις ε, που έγιναν για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης, εμείς ε, στην Επιτροπή DCI συζητήσαμε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή DCI συμφώνησε να τροποποιήσει το κείμενο. Έτσι λοιπόν πράξαμε έτσι όπως ζητήθηκε από την ομάδα εργασίας. Είναι και ο συνάδελφός μου εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο για να απαντήσει στα θέματα που αφορούν την Λατινική Αμερική. Ο συνάδελφος από τη ΓΑΜΑ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να τονίσω ορισμένα σημεία που τέθηκαν. Καταρχήν ευχαριστώ τις ομάδες εργασίας για τη συνεργασία τους και ε, για το έργο που επιτέλεσαν ε, μαζί μας. Λαμβάνουμε υπόψη τα σχόλια που υπόθηκαν. Εμείς σκοπεύουμε να τα λάβουμε υπόψη κυρίως ό,τι αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Έτσι, λοιπόν, όταν γίνονται αφορές στις ομάδες στόχου ή στους δείκτες, την ανάγκη δικτών, αυτό θα το διευκρινίσουμε περισσότερο όταν έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα που τίθενται σε εφαρμογή και αιτήσια προγράμματα που τίθενται σε εφαρμογή. Η Κομισιόν θα έχει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά όταν θα ασκεί το ε, δικαίωμα πρόσβαση δημοκρατίας. Ε, να αναφερθώ τώρα στην ανακούφιση της φτώχεια, πάνω από το 40% πόσο κάνουμε στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας Λατινικής Αμερικής αφιερώνεται στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής ε, σε ορισμένε περιπτώσει μέσω προγραμμάτων για την άμβληση της φτώχεια. ορισμένες φορές μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά τώρα το νέο μέσο, το Latin American Investment Facility, θα ήθελα να σας πω ότι θα θέλαμε το μέσο να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή και θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι έγινε πολύ σημαντική προσπάθεια στα έγγραφα της ενδιάμεσης αναθεώρησης ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών. Ίσως να μην κάνουμε αρκετά, αλλά εμείς ε, έχουμε ε, ουσιαστικά κάποια κονδύλια προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Θα το πράξουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Τώρα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στήριξη θα το συζητήσουμε και πάλι στην Επιτροπή αυτή ε, να μην ε, ξεχνάμε σε ό,τι αφορά την ε, τριγωνική συνεργασία. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος. Δηλαδή θέλουμε σε αυτό να συμμετέχουν όλες οι χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεδομένου ότι εγκρίναμε τα έγγραφα αυτά, έχει ολοκληρωθεί η δουλειά του Κοινοβουλίου επί των εγγράφων αυτών. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τις προθεσμίες. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Θεοχάρους για τη μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό σε μισή ώρα. Ξέρω ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη, έκθεση και θα ήθελα να δώσω το λόγο της αμέσως στην κυρία Θεοχάρους. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στον Τόμ Μόργαν ε, για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης, όπως επίσης στον κύριο Πολοσόφ και στους συναδέλφους τους Σκιώδη, συζητητές Νόιζερ, Κλίντς, Λέβι, Ντέβα και Τσίμερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε όχι μόνο στην ανακούφιση της ε, φτώχειας, ε, αλλά κυρίως στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι αυτή η γενικότερη φιλοσοφία μας και αυτή ήταν από την αρχή. Θέλαμε από την αρχή να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη σημασία των ε, εξή παραμέτρων. Πρώτον, ένα περιβάλλον σταθερό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ένα νομικό πλαίσιο χωρίς διαφθορά, το γεγονός ότι η βιομηχανοποίηση οδηγεί σε οικονομική κρίση και σε κλιματική αλλαγή. Επίσης, ε, εκπαίδευση σε θέματα υγείας επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στους ε, παράγοντες αυτούς, ε, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού για τον τομέα της υγείας σε, χώρες, σε αυτές τις χώρες, όπως επίσης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, ποιοτική και Αντιμετωπίσαμε επίσης και το θέμα το, της χαμηλής εκπροσώπησης των ε, ε, χωρών των φτωχότερων στη, στα διεθνή φόρα. Πρώτον, έχουμε τις προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες και δεύτερον, οι προκλήσεις για τις χώρες δωρητές. Η πρώτη πρόκληση έχει να κάνει με την οικονομία. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα έπρεπε να φορτώνουν τις επιχειρήσεις με πάρα πολύ γραφειοκρατία. Τα Επίσης πρέπει να προωθήσουμε πρόσβαση των, πιστώσεων, πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ε, πιστώσεις. Ε, επίσης να τους δώσουμε να δώσουμε στους φτωχότερους τη δυνατότητα ιδιοκτησίας της γης τους. Επίσης, οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα έπρεπε να εφαρμόσουν ε, την ε, σύμβαση κατά της διαφοράς. Επίσης, ανεξάρτητη, ανεξάρτητα κοινοβούλια για καλύτερη δημοκρατία και κάτι ακόμη ενισχυμένη και καλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Όσον αφορά τις ε, κοινέ προκλήσεις, ε, θα έπρεπε 20% ε, της εθνικής και της ευρωπαϊκής βοήθειας να αφορά την εκπαίδευση για θέματα υγείας, ενθάρρυνση των τοπικών γιατρών και άλλων επαγγελματιών του τομέα, να ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο της κοινότητάς τους, μεγαλύτερη έμφαση για την ιατρική φροντίδα, ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους, επένδυση επένδυσης στις πράσινες θέσεις απασχόλησης ε, και συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους όσον αφορά του, τις προκλήσεις για τους δωρητές. Έχουμε επίσης τρία ακόμη κεφάλαια που αφορούν ε, την ε, βοήθεια. Πρέπει να τηρούνται υποσχέσεις υποστήριξης, πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, τηρήσει τις υποσχέσεις της σε εμπορικό επίπεδο, να απλοποιήσει το σύστημα ενίσχυσης και να επενδύσει ευφιέστερα ε, στην, ε, στην εκπαίδευση των πολιτών. Όσον αφορά το G20, να καταργηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι και θα έπρεπε η G, η ομάδα των G20 να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα αυτό όσον αφορά τη δημιουργία υποδομών. Πρέπει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του τομείς ε, που είναι επωφελεί για τις χώρε εταίρου, ε, ε, όπως για παράδειγμα οι οικονομικοί τομεί που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και στον τομέα τον εκπαιδευτικό επίση. Πρέπει οι φοιτητέ, ακόμη και όταν σπουδάζουν στο εξωτερικό, να επιστρέφουν στις χώρε του και να ασκούν το επάγγελμά του εκεί. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόζει κριτήρια ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως επίσης ε, και να είναι πιο στοχευμένη η ενίσχυση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει καλά προγράμματα παρατήρησης των εκλογών για καλύτερη δημοκρατική εκπροσώπηση σε παγκόσμιους, σε παγκόσμιους τους ε, οργανισμούς. Αυτά λοιπόν και περιμένουμε τις ε, προτάσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα κάποιες ε, Ευχαριστώ την κυρία Θεοχάρους για αυτή τη σύνοψη της ε, έκθεσής σας, Κρυσνέσερ και τα μέλη της ΑΣΕΝΤΗ φυσικά συμφωνούν ε, στο ότι επικεντρώνεστε στο θέμα των θέσεων, ε, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και σε όλες τις πτυχές που αφορούν την κατάργηση της γραφειοκρατίας, της μικρές και μεσές επιχειρήσεις, πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά επίσης ε, και το να διευθυνθεί το θέμα της ιδιοκτησίας της ε, γης. Κατά ε, αντιμετώπιση της διαφθοράς, να προωθήσουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί και μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες το να ε, δημιουργηθούν αξιοπρεπεί θέσει εργασία είναι ο μόνο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει ε, τι αναπτυσσόμενε χώρε να βγουν από τη φτώχεια. Εμεί θα πρέπει να προσφέρουμε όσο το δυνατόν ένα πιο σταθερό περιβάλλον για να μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιε θέσει εργασία και η ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία του ΔΟΕ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ που το αναφέρετε. Ε, εμείς θεωρούμε ότι εδώ. Υπάρχει όμως ε, κατά κάποιο τρόπο γίνεται μια σύνοψη της ε, ε, συνένεσης για την ανάπτυξη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να διαφωνήσει. ήταν πολύ δύσκολο. Αυτά που λέτε εδώ είναι πολύ ευρεία. Εμείς θέλουμε να περιοριστούμε σε κάποιες τροποποιήσεις λόγου χάρη για την παιδική εργασία. περιοριζόμαστε όμως αυτά τα μικρά σημεία γιατί γενικά συμφωνούμε μαζί σας επί του συνόλου σας. Ευχαριστώ πολύ.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 τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τις ε, παρουσιάσει κανείς ε, με τη μορφή μιας περίληψης. Ε, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την έκθεση, αλλά πρέπει να διερωτηθεί κατά πόσον παρόλα αυτά θα πρέπει να έχει το θάρρος να κάνει κάποιες ερωτήσεις επί τη ουσία Οι ερωτήσεις αυτές να είναι πρόκληση, προκλητικές και στη διατύπωσή τους και στο στόχο τους. Γιατί ένα πράγμα πρέπει να διαπιστώσουμε, παρότι η κατάσταση σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Αφρική, εξακολουθεί να είναι ανικανοποιητική, το θέμα δεν είναι ότι δίδονται λίγα ή πολύ λίγα χρήματα. Όχι, τα τελευταία 50 χρόνια δόθηκαν αρκετά κονδύλια, δισεκατομμύρια κονδυλίων. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια διέθεσε 2,5 δις ευρώ. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα στο σύνολό του δεν είναι ικανοποιητικό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διερωτηθούμε, μα τι δεν πάει καλά. Αν δούμε λοιπόν λιγάκι όλο τον πλανήτη και σε όλες τις υπήρους ε, υπήρξαν και υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σε ορισμένες υπήρους κατέστη δυνατόν τουλάχιστον ε, ε, σε μεγάλο βαθμό οι χώρες να προχωρήσουν στην Ασία, στην Ασία σίγουρα και στη Νότια Αμερική χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο. Η Βραζιλία είναι η, Αργενία, η Αργεντινή ήτανε, τώρα πια δεν είναι. Πάντως στην Αφρική κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Η συγγήτρια πολύ σωστά λέει αυτό οφείλεται στη διαφθορά, στη φοροδιαφυγή. Δικαίως ε, αναφέρεται σε φαινόμενα όπως παιδική εργασία και ούτω καθεξής. Όμως ε, αυτά είναι ε, τμηματικές παρατηρήσεις σε γενικές γραμμές, κατ' ουσίαν, δεν έχουμε λειτουργούντα, εύρυθμα λειτουργούντα κράτη. Δεν είναι κράτη όπου ε, να μπορεί κανείς να μιλάει για σταθερή διακυβέρνηση. Στις χώρες αυτές επικρατούν η παραοικονομία, η διαφθορά και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι οποτεδήποτε ξεσπάει πόλεμος ξαφνικά υπάρχουν χρήματα. Όταν όμως ε, τελειώνει η πόλεμη και ελπίζει κανείς ότι εφόσον υπάρχουν χρήματα, άρα θα μπορεί η κοινωνία των πολιτών να δραστηριοποιηθεί, τότε ξαφνικά τα χρήματα κάπου χάνονται σε κανάλια που δεν γνωρίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς οφείλουμε να διερωτηθούμε το εξής. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να καταστήσουμε δυνατό τον έλεγχο, τον καλύτερο έλεγχο, να ελέγχουμε καλύτερα τους ε, αποδέκτες και να διασφαλίζουμε ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως ε, στόχο, επειδή είμαι αισιόδοξο το λέω, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι μια ανοιχτή, αλλά με την πάροδο των ετών θα πρέπει να, ε, ιδρυθεί, να ιδρυθούν κοινωνίες με βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο. Δηλαδή κοινωνίες που να βασίζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνίες όπου ε, το περιβάλλον δεν καταστρέφεται, αλλά οι φυσικοί πόροι προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Και επίσης σε μια κοινωνία όπου υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά είναι οι αρχές της Ευρώπης. Οικονομία, οικολογία και κοινωνικά θέματα. Αυτή πρέπει να είναι η στόχη μας. Και αυτό που κάναμε είναι το εξής. Δώσαμε εδώ και εκεί κάποια χρήματα, αλλά γενικά όμως ε, τη σφαιρική προσέγγιση δεν την ε, προαγάγαμε επιτυχώς. Βεβαίως ε, και εμείς αντιφάσκουμε. Από τη μια ανοίγουμε το πορτοφόλι μας και είμαστε γενναιόδοροι. Όταν όμως έρχονται οι χώρες ε, και λένε θέλουμε εμείς να σας εξάγουμε αυτό που μπορούμε, δηλαδή γεωργικά προϊόντα, τότε τους λέμε και εμείς, α, ξέρετε κάτι δεν γίνεται, οι τιμές σας είναι πολύ χαμηλές, πρέπει και εμείς να ορίσουμε τιμή κατόφλι για να μην καταστρέψουμε την οικονομία μας. Αυτό όμως δεν γίνεται, είναι ασυνεπές. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το επισημάνουμε με κάθε παρησία και να έχουμε κατά νου και κάτι άλλο. Τώρα, κατά πόσο ισχύει αυτό ή όχι. Εγώ δεν το μπορώ να το πω γιατί δεν είμαι εμπειρογνώμων, αλλά ο συνάδελφός μου, κύριος Χέρενς, μου επισήμανε ότι στο Παρίσι, τελειώνω, υπάρχει μία λέσχη της Σαχάρας που ασχολείται με την αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτή λοιπόν η λέσχη κατέληξε, πολύ ενδιαφέρον αυτό, στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν τελικά δεν περάσει μια χώρα τη βάση της εκβιομηχάνησης. Όχι ότι πρέπει κανείς παντού να κατασκευάσει χαλιβουργία, βιομηχανία χαλιβουργίας, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια βιομηχανία. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε αυτομάτως από τη γεωργική κοινωνία στην κοινωνία των υπηρεσιών. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να ξέρουμε ποια είναι τα απαραίτητα βήματα. Γιατί οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι σωστό. Εμείς δεν διαφωνούμε με την έκθεση, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα επί τη ουσία και αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Ευχαριστώ, κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια παράθεση. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο συγγραφέας. Πρόκειται για μία παράθεση προέρχεται από μία συνέντευξη που είχαμε έναν αρχηγό Αφρικανικού κράτους ε, μου είπε ότι είναι το κράτος μου διεφθαρμένο γιατί είναι οι υπάλληλοι μου διεφθαρμένοι, είναι διεφθαρμένοι γιατί τους πληρώνω, ε, τους κακοπληρώνω, γιατί δεν υπάρχει ε, τίποτα στο Ταμείο του Κράτους, δεν υπάρχει το Ταμείο του Κράτους γιατί δεν πληρώνουν τους φόρους οι φορολογούμενοι, δεν πληρώνουν τους φόρους οι φορολογούμενοι γιατί κανείς δεν έρχεται να επενδύσει στη χώρα μου και τελικά αν έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα μου, θα μου πει «Α, θα έρθω να επενδύσω μόλις πάψει να είναι διεφθαρμένη η χώρα μου». Και μου λέει, «Ε, βοηθήστε με να μετατρέψω αυτό το φαύλο κύκλο σε ένα κύκλο αρετή. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη μικρή ιστορία βρίσκεται όλο το νόημα της κατάστασης. Ε, ε, ουσιαστικά μου αποκάλυψε την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κράτος του. Ε, θα μπορούσα να αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα για να υπογραμμίσω εδώ το παράλογο της κατάστασης στην ακτή του Παραδείγματο χάρη, ο Μπάγκο βρίσκει χρήματα ε, για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, αλλά όχι υπό τη μορφή φόρων. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει μια δυνατότητα συλλογής ε, κονδυλίων για την ανάπτυξη. Εμείς τα τελευταία 25 χρόνια ε, μου είπε ότι προσπαθούμε να ε, συλλέξουμε το 25% των ε, φόρων και φυσικά χρειάζονται να γίνουν δράσεις για την καταπολέμηση του AIDS γιατί κανείς δεν μιλάει σήμερα γι' αυτό ή για το υγειονομικό τομέα κανείς δεν μιλάει σήμερα γι' αυτό πρέπει λοιπόν να βρούμε χρήματα και γι' αυτά και όχι μόνο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στις αφρικανικές χώρες και η η ακτή του ελεφαντοστού, ξέρετε ότι είχε ένα ε, ποσοστό ανάπτυξη συνεπέ και βλέπουμε τώρα να πιστοχωρεί. Πρέπει να αναρωτηθούμε. Ο κύριο ε, Κλίνς τώρα ανέφερε το εξή. Στην Αφρική υπάρχει μια πολύ διαφορετική κατάσταση σήμερα σε σχέση με τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μονίμως τον ίδιο Πάνω από το ίμιση ε, των ε, κατοίκων ζουν στις πόλεις δεν ε, έχουν εργασία. Υπάρχει λοιπόν μια κοινωνική έκρηξη η οποία βρίσκεται ενώπιόν μας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε ένα στάδιο εκβιομηχάνησης, δηλαδή να μετατρέψουμε τον πλούτο επιτόπου και να υπάρξει προστιθέμενη αξία για τους ε, πολίτες. Ο στόχος της ε, ανάπτυξης ε, είναι να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία αυτή η ανάπτυξη για να μπορεί η ίδια η χώρα να στηρίζει τον εαυτό της. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ νομίζω ότι εντάξει εδώ έχετε βρει μια φόρμουλα, δεν μπορούμε να αντιταχθούμε, αλλά νομίζω πρέπει να πάμε λίγο πιο μακριά να ρωτηθούμε για τον αντίκτυπο της Κίνας. Πάντοτε λέμε, ναι, υπάρχουν ε, τρόφιμα και τα λοιπά, υπάρχουν πολλά θετικά και αρνητικά, όμως εγώ θεωρώ απαράδεκτο μια χώρα να φτάσει να ανταγωνίζεται την ε, οικονομία. και αυτό φυσικά έχει να κάνει με το πόσο χαμηλό είναι το νόμισμα της Κίνας και έτσι μπορούν να προβαίνουν σε ένα εμπορικό dumping. Και αν δούμε και τους κανόνες ε, του ΠΟΕ, δεν βρίσκουμε ε, επαρκή επιχειρήματα για να τους καταδικάσουμε επειδή κάνουν αυτό το εμπορικό dumping. και ουσιαστικά έχουν ένα τόσο δύναμο νόμισμα που μπορούν να προβαίνουν σε αυτό το εμπορικό dumping. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στο κατάλληλο πλαίσιο. Και θα ήθελα να κλείσω όμω και με κάτι θετικό όλα σε λέω για τη διακυβέρνηση. Δυστυχώ είναι αλήθεια. Αλλά αν ε, είχαμε κάνει μια διαπίστωση πριν 30 χρόνια, η διαπίστωση θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Υπήρξε πρόοδος, ε, η Μοζαμβίκη τα πηγαίνει αρκετά καλά και είναι μία από τις ε, λίγες χώρες η οποία ουσιαστικά πληρεί τους στόχους της χιλιετίας γιατί ακριβώς περνά από μια φάση εκβιομηχάνηση και υπάρχει και μια προσθέμενη αξία που έχει δημιουργηθεί επί τόπου. Εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να δούμε και πρέπει να ρωτηθούμε και για το πώ αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα τη φτώχεια, πώ το προσεγγίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να εντοπίσουμε κάποια σημαντικά think tank που να μπορούν να μα δώσουν τα επαρκή επιστημονικά επιχειρήματα για να διατυπώσουμε και εμεί τις απαντήσεις μας. Γιατί ο κόσμο είναι γεμάτο γκουρού, γεμάτο ανθρώπου που λέει «Α, αυτό πρέπει, το τάδε ή το δίνα». Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να δείχνουμε εδώ μια τεχνική προσέγγιση στην ανάλυση μας. Επίσης, είδα ότι αναφερθήκατε και στο πρόβλημα της υγείας. Παραμένει ε, ε, ε, ο υγειονομικός ένας τομέας που πρέπει να επικεντρωθούμε και έχουμε και το πρόβλημα και των γιατρών και της φυγής εγκεφάλων. Εγώ νομίζω ότι σε μια καλή σχέση βορρά-νότου θα μπορέσουμε να εξεύρουμε λύσεις. Ε, Παίρνουμε χάρη να δίνουμε ε, υποτροφίες ε, σε Αφρικανούς φοιτητές, οι οποίοι θα έπρεπε να δέχονται χάρη σε αυτές τις υποτροφίες να θέτουν ουσιαστικά την γνώση τους την υπηρεσία της χώρας προέλευσής τους δεν ε, είναι λογικό να έχουμε τελικά ε, ένα πολύ μεγάλο αριθμό γιατρών που να έχουν καταρτιστεί σε μια χώρα και τελικά στη διάθεση της χώρας ε, να μένουν ελάχιστοι. Αντί να μιλάμε λοιπόν για μηδενική μετανάστευση, θα πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα και να δίνουμε λόγου χάρη πολλαπλές θεωρήσεις λόγου χάρη στην, σε φοιτητές οι οποίοι να μπορούν να ωφελούν τους συμπολίτες τους στη χώρα προέλευσής τους με τις γνώσεις που αποκτούν. Εγώ νομίζω ότι η έκθεση είναι καλή, αλλά αξίζει να κάνουμε μία βάθος σε συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα που θέτονται. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Έτσι λοιπόν σας ζητώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχήν ε, για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και για την ε, προσπάθεια το, να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορώ βέβαια να καταλάβω πάρα πολύ καλά γιατί προβάλλονται ορισμένα αιτήματα. Ο συνάδελφος κύριος Κλίνς, αλλά και εσείς το εξηγήσατε. Πιστεύω όμως παρόλα αυτά ότι είναι αισθητό το ότι το ενδιαφέρον για το θέμα της φτώχειας, που καταρχήν υποτίθεται δεν θα περιλαμβανόταν καν μέσα στην έκθεση, προέκυψε μετά από το ενδιαφέρον των συντονιστών. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα αυτό λιγάκι χάνει τη σημασία του. Ε, μεγαλύτερη σημασία αποκτά το ε, πώς ε, μπορεί κανείς στο μέλλον να μιλήσει καλύτερα για τη συνεργασία, για τις θέσεις εργασίας, όμως ε, το θέμα του πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, αυτό μοιάζει δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο, κυρίως ε, εμείς ε, ως Επιτροπή Ανάπτυξης, να ασχοληθούμε με αυτά τα οποία έγιναν το Φεβρουάριο στα Ηνωμένα Έθνη. Κυρίως εκεί που γίνεται λόγος ε, για την ε, έκθεση περί κοινωνικής κατάστασης ανά τον κόσμο. Εξάλλου, ε, φάνηκε ότι το θέμα της φτώχειας πρέπει να αναθεωρηθεί. Ναι, μεν, τα τελευταία χρόνια κατέστη δυνατόν σε, αρκετούς, σε αρκετές περιφέρειες της χώρας αρκετά σημεία να περιστεί η φτώχεια, αλλά στην υποσαχάρη Αφρική και σε άλλες περιοχές του κόσμου συνέβη το αντίθετο. Αυξήθηκε η φτώχεια. Και έτσι λοιπόν οι στόχοι της χιλιετίας μοιάζουν να κινδυνεύουν. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλες προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να είμαστε συντομότεροι, πιο, να είναι πιο ευσύνοπτο το κείμενο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το θέμα της φτώχειας πρέπει να αφαιρεθεί. Εφόσον παραμένει λοιπόν το θέμα της φτώχειας, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθούμε περαιτέρω και χρειαζόμαστε και μία συζήτηση για το ότι το 80% του ε, παγκόσμιου πληθυσμού δεν ε, απολαμβάνει κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση. Το 80%. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε το πώς ακριβώς αυτό το θέμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι σημαντικό κυρίως για εμάς τους Ευρωπαίους. Αυτό το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που μπορεί κανείς να θίξει. Εμένα, ξέρετε, μου μοιάζει λιγάκι ότι τα θέματα που αφορούν στην κριτική κατά της κακής διακυβέρνησης, ε, της ε, διαφθοράς, αυτά κατά κάποιον τρόπο αποδίδονται στις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες, στο ότι είναι υπανάπτυκτες, στο ότι εν μέρη υπάρχουν ε, απαράδεκτες ε, οικολογικές ε, συνθήκες. Αυτό δεν έχει άμεσα σχέση με την κακή διακυβέρνηση, έχει σχέση και με τις δικές μας τις ενέργειες ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη. Δηλαδή ενδιαφερόμαστε περισσότερο να συμμετέχουμε οικονομικά, να κάνουμε επενδύσεις. Αυτό είναι αυτονόητο. Όμως, ε, κάνω το ερώτημα, γιατί ας πούμε η Κίνα αυτή τη στιγμή προηγείται τόσο πολύ των Αφρικανικών κρατών. Στην Αγγόλα το είδαμε την πήραμε την απάντηση. Ξέρετε γιατί, διότι οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται μόνο για τους πόρους, αλλά ενδιαφέρονται και στο να υποβάλουν συγκεκριμένε προτάσεις για την ανάπτυξη υποδομής. Και πάμε στο επόμενο θέμα, που κατά την άποψή μου πρέπει να προβληθεί περισσότερο στην έκθεση. Μία απάντηση που δόθηκε ήταν ότι ε, σε αυτά τα μεγάλα προγράμματα συμμετέχουν σχεδόν αποκλειστικά Κινέζοι εργαζόμενοι και ότι οι κάτοικοι της ε, δεν μπορούν να συμμετάσχουν γιατί το 80% είναι αναλφάβητοι έτσι και αλλιώ. Άρα δηλαδή τι πρέπει κανεί να κάνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Γερμανία ε, να απευθυνθούν στην Αγκόλα και η Αγκόλα να ζητήσει από τη Γερμανία και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπαίδευση, να εκπαιδευτούν. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο πανεπιστήμια, να πάμε πιο κάτω χρειαζόμαστε κυρίως ε, στην εκπαίδευση εξειδικευμένων εργαζομένων μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε πολλά άλλα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς με τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να φέρουμε έτσι κάποια ισορροπία, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το βάρος αυτής της έκθεσης, κυρίως όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ξέρετε, θα καταθέσουμε ε, την δέουσα, τον δέοντα αριθμό τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοχάρους, για την έκθεση αυτή. Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα αν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της φτώχειας και της ε, ανεργίας, δεν θα χρειαζόμασταν την Επιτροπή αυτή. Οπότε αυτό όλοι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Δεν συμφωνώ απολύτως με όλα τα σημεία. Για παράδειγμα, στο σημείο που λέτε ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον ε, σημαίνει περισσότερες θέσεις απασχόλησης και έναν πιο ασφαλή και βιώσιμο τρόπο καταπολέμησης της φτώχειας. Πολύ καλή δήλωση, αλλά τι ακριβώς θα πει η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και ποιος ακριβώς θα πλουτίσει και τι ακριβώς σημαίνει φτώχεια εν Μπορεί να έχει κανείς ένα καλό επιχειρηματικό πλαίσιο που έχει ως αποτέλεσμα οι δυτικέ χώρες να επενδύουν. Αλλά μπορεί αυτό να μην οδηγήσει σε μεγαλύτερο πλούτο για ολόκληρη τη χώρα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα, μπορεί ηλεκτρονικά απόβλητα να χρησιμοποιούν από τις ε, ανεπτυγμένες χώρες. Πώς ακριβώς λοιπόν γίνεται αυτό, πώς ακριβώς θα, είμαστε θα είναι εποφελής η κατάσταση για τον πληθυσμό στο σύνολό του. Από απόψεως φυσικών πόρων η Αφρική είναι μία από τις πλουσιότερες υπήρους στον κόσμο και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι χώρες αυτές πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν και να επεξεργαστούν ε, τις πρώτες ύλες τους. Δεν θα είναι ανάγκη, να ε, πουλούν ψάρια ε, στους Ευρωπαίους αλληλείς. Το θέμα της εμπορικής πολιτικής είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με τους αναπτυξιακούς ε, στόχους της καταπολέμησης της φτώχειας. Κάτι ακόμη που πιστεύω ότι λείπει είναι μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το μέλλον όλων μας και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι θα ήταν κρίμα οι αναπτυσσόμενες χώρες να επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν οι ανεπτυγμένες χώρες καταστρέφοντας τους φυσικούς πόρους και καταστρέφοντας το περιβάλλον. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε μία προσέγγιση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια, που μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν μιλάμε για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά, τηλέφωνα, να μην χρειάζεται δηλαδή να εξαφανίζονται τα δάση για να μπορούν να έχουν καύσιμα οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει λοιπόν στην πράσινη ανάπτυξη να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη έμφαση και είναι κάτι που χρειάζεται σε όλο τον κόσμο και είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ουσιαστική σημασία. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχουμε μία πολιτική που μειώνει τις ευκαιρίες απασχόλησης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες όταν εξάγουμε κοτόπουλα για παράδειγμα που κανένας Ευρωπαίος καταναλωτής δεν θα ήθελε να αγοράσει και έτσι πολύ, απλώς, ε, πολύ απλά το προωθούμε στις αφρικανικές χώρες ε, κοτόπουλα που δεν θέλουμε τα στέλνουμε στο Καμερούν Και το ίδιο ισχύει και για την αλληλευτική μας πολιτική, όπου ανταγωνιζόμαστε με τους ντόπιου αλληλείς σε χώρες όπως η Σενεγάλη, η Γουινέα Μπισάου, Μαυριτανία, 600.000 άνθρωποι έχουν ε, επηρεαστεί από τον ε, αλλιευτικό τομέα λόγω της κατάστασης αυτής και έχουμε πάρα πολύ αφαιρέσει θέσεις απασχόλησης αντί να δημιουργήσουμε. Επομένω πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στο πλαίσιο της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεβίν για τα σχόλια αυτά. ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριος Ταμάς Φαρνή ή κυρία Νικολέτα Μέρλου. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι παρόν. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε και για την ε, πολύ φιλόδοξη και πλήρη έκθεση. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή, οπότε έχουμε κρίση, όμως βέβαια τα θέματα της μείωσης της φτώχειας δεν πρέπει να προβάλλονται μόνο σε στιγμές κρίσης. Όπως ανέφεραν και ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την τελευταία δεκαετία είχαμε πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική, όμως ε, αυτό δεν μεταφράστηκε σε βελτίωση στο κοινωνικό επίπεδο, ούτε στην ε, επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και η κρίση ήρθε τώρα να διακυβεύσει ε, να, ε, και μια ακόμη φορά τα επιτεύγματα των χωρών αυτών ως προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Ε, φυσικά πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική προστασία και χαίρομαι που ανέφερε η κυρία Τζίμερ ε, το θέμα της κοινωνικής προστασίας ε, και οι δύο πολιτικές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για να μετριάσουν τα αρνητικά αποτελέσματα της κρίσης και για την αύξηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν δύναμε, θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την έκθεση όταν ε, ορίζετε τη φτώχεια, ίσως ε, να θέλετε να πάτε παραπέρα από την ε, φτώχεια που αφορά την έλλειψη εισοδήματο, να αναφερθείτε και στον κοινωνικό αποκλεισμό και σε άλλα στοιχεία. Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι αναφέρεστε στην ε, ατζέντα για ε, την αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ, αλλά ίσως θα ήταν καλό να αναφέρεστε και στο ε, Global Jobs Pact που υιοθετήθηκε πέρσι από τη ΔΟΕ. Δεν το είδα να αναφέρετε. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε σαφή συνδεσμό μεταξύ των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης. Και εδώ αναφέρουμε στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Αυτά είναι γενικά σχόλια, αλλά εμείς από την πλευρά της Κομισιόν εξετάσαμε τις παραγράφους της έκθεσης και κάναμε λεπτομερή σχόλια. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι σήμερα έχουμε χρόνο να τα αναφέρουμε εδώ. Αλλά ευχαρίστως να στείλω αυτά τα σχόλια γραπτό στην εισηγήτρια και στην γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θοχάρους έχει το λόγο για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις πολύ επικοδομητικές ε, παρατηρήσεις τους. Δεν διαφωνώ με καμιά. Εδώ καταθέσαμε μια γενικότερη πολιτική. Ήθελα να σας θυμίσω ότι ο Μάρκ Τουέν στο βιβλίο του «Ο του βασιλιά Λεοπόλδου» εκεί στην εισαγωγή λέει κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να απολογηθώ μπροστά σε κάθε Αφρικανό κάθε φορά που φτάνω στην Αφρική. Δεν θα σας το πω, γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά όποιος θέλει μπορεί να βρει το βιβλίο και να το διαβάσει. Σε αυτή την έκδοση που έχω στα χέρια μου λέει ακόμη ότι όταν το Κονγκό έγινε ανεξάρτητη χώρα, είχε 17 εκατομμύρια πληθυσμό και 17 τυχιούχους πανεπιστημίου. 17 πανεπιστημίου. Γι' αυτό και ιδρύθηκε αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Λουμούμπα στη Μόσχα που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανάπτυξη των Αφρικανικών κρατών. Όλα τα μέτρα που έχετε εισηγηθεί είναι πολύ σωστά και περιλαμβάνονται στο report εκτός από το, την χρήση των think tanks για την επεξεργασία των οδηγιών αυτών αλλά ως γενικότερη πολιτική νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να πω ότι η κακοποίηση των Αφρικανικών κρατών συνεχίζεται και έχετε δώσει όλοι πολλά παραδείγματα για το πώς εξακολουθούμε να το κάνουμε στην Ευρώπη αυτό το, αυτό το θέμα. Η, το exploitation, το, το, το commercial exploitation. Τώρα, όσον αφορά ένα ζήτημα αν θα πρέπει πρώτα να εκδημοκρατικοποιηθούν αυτές οι χώρες και στη συνέχεια να δούμε την πρόοδο και την ανάπτυξη ή αν παράλληλα μπορούν να γίνουν αυτά τα δυο, ναι αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο εισηγούμαστε την παρέμβαση προς την κοινότητα. Εγώ δεν έχω εισηγηθεί να δίνουμε χρήματα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θα αναπτυχθεί η Αφρική και ο τρίτος κόσμος ή ο underdeveloped κόσμος. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτή την προσέγγιση που θα αναστείλει, θα περιορίσει και το μεταναστευτικό ρεύμα και θα κρατήσει τους ανθρώπους στον τόπο τους. Η παρέμβαση προς την κοινότητα. Το έχω πει από την πρώτη συνάντηση. Βεβαίως όλα θα τα λάβουμε υπόψη και τις εισηγήσεις και σας ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι ευγνώμων για αυτά που έχετε πει. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι Παρασκευή 26 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας σήμερα θα εξεταστεί και κλεισμένων των θυρών. Καλό όλους όσους ε, δεν είναι σε εξής κατηγορίες να αποχωρήσουν. Βοηθή... Ε, ευρωβουλευτών, ευρωβουλευτές, ε, υπάλληλοι πολιτικών ομάδων και υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη της Γραμματείας βέβαια. Παρακαλώ οι κλητήρες ε, να ελέγξουν ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από εδώ και στο εξής και